Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ακόμη και αν δεν έχουν έρθει τόσο πολύ, Αλλά 9 η ώρα σημαίνει 9 η ώρα. Έχουμε μία ομάδα ε, επισκεπτών των Deep Halls, τους καλωσορίζω στη συνεδρίασή μας. Και τώρα, να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση είναι δημόσια και επίσης μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά στο ίντερνετ. Πρώτο θέμα της μέρης διάταξης είναι η έγκριση της μέρης διάταξης. Υπάρχουν προτάσεις τροποποίησης της. Όχι. Ωραία. Να τονίσω ότι η κυρία Μόσκα μας παρακάλεσε να αντιστρέψουμε τα σημεία 8 και 9. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε, οπότε το εγκρίνουμε. Επαναλαμβάνω, το 8 και 9 θα αντιστραφούν. 2. Έγκριση των πρακτικών. Ως συνήθως, εάν μέχρι τέλους της ε, συνεδρίασης. Δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις τροποποίησης, θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Οπότε περνάμε στο 3. Ανακοινώσει του Προέδρου. Ως συνήθως έχετε ένα κατάλογο των ε, επιστολών που έχουν αποσταλεί Και αν θέλετε να δείτε το περιεχόμενο κάποιες επιστολής, ζητήστε το από τη γραμματεία. Αναφέρθηκα ότι λοιπόν υπάρχει web streaming. Είναι δυνατό λοιπόν μέσω του διαδικτύου να μας παρακολουθήσει ολόκληρος ο κόσμος. Να το έχετε υπόψη σας. Και Παρακαλώ να βοηθήσετε τους διερμηνείς ε, να μιλάτε σαφώς και όχι πολύ γρήγορα για να μπορούν να αποδίδουν επακριβώς αυτά που λέτε. Κάποιες ε, εξελίξεις της ε, διαπραγματεύσεις για εμπορικά θέματα, ο δέκατος γύρος διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία έλαβε χώρα μεταξύ 22 και 29 Απριλίου οι συζητήσεις ε, είναι πολλά υποσχόμενες. Αναφέρθηκαν όλα τα σημαντικά θέματα, δασμοί, δημόσιες προμήθειες, σιδεροδρομικός τομέας και γεωγραφικές ενδείξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί μια κάποια δυναμική σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Οπότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπογραφεί συμφωνία με την Ιαπωνία. Θα υπάρξει περαιτέρω πρόοδος εν ώψη της συνάντησης κορυφής Ένωσης Ιαπωνίας που θα έχουμε το Μάριο. Επίσης, για τη διαπραγματεύσεις για τα πράσινα προϊόντα, green goods, στα πλαίσια του ΠΟΕ, η διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα φέτος, ε, συγγνώμη, τώρα, 4 με 6 Μαΐου και αφορά κυρίως τον κατάλογο των πρασίνων προϊόντων. Η Επιτροπή το ζήτησε μαζί μας 16 Απριλίου. Οι εξελίξεις για το TTIP φυσικά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Οι εισηγητές White and Hedge στη Γερουσία και Paul Wine στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν υποβάλει προτάσεις που εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές αλλά τώρα στην Ολομέλεια της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ προκαλούν ευρύτερες συζητήσεις και φαίνεται ότι υπάρχει πλειοψηφία για αυτή την αρχή πρόθεση του εμπορίου, Trade Promotion Authority. Υπάρχει πλειοψηφία λοιπόν στη Γερουσία αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Διότι το Ρεπουμπλικάνικο κόμμα έχει πολλές επιφυλάξεις. Λέγεται ότι 75 αντιπρόσωποι δεν θα ψηφίσουν ενώ από πλευρά των Δημοκρατών είναι μόνο 15 υπέρ, οπότε δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα υπάρξει πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Πολιτειών. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε. Να δούμε αν τουλάχιστον θα αναβληθεί η ψηφοφορία ούτω ώστε να γίνουν περαιτέρω διαβουλεύσεις κατά το Σαββατοκύριακο. Εάν αποφασιστεί αυτή η αρχή, λοιπόν, θα υπάρχουν τρία τμήματα. Ένα θέμα για τις ε, συνθήκες εμπορίου, ένα για τη διαφάνεια και ένα τρίτον για τα διαδικαστικά θέματα. Και ο δεύτερος λοιπόν πυλώνας είναι πολύ σημαντικός γιατί εκεί θέτει το Κογκρέσο προϋποθέσεις για τη διαφάνεια που εμείς υποδειγματικά τις έχουμε εκπληρώσει όσον αφορά για παράδειγμα τα έγγραφα και το Κογκρέσο θέλει και μια τέτοια ομάδα επίβλεψης ε, που εμείς την έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Αυτή η αρχή θα έχει περιορισμένη εντολή μέχρι την πρώτη Εβδόμου 18 για να υπάρχει επαρκής χώρος για διαπραγματεύσεις. Αν δεν επιτύχουμε μέχρι τέλους του έτους να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αλλά δεν νομίζω ότι με βάση της, ε, τη συγκυρία τώρα είναι πολύ πιθανό αυτό. θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά την κατάσταση και ξέρετε ότι κυρίως προσπαθούν να επικυρώσουν τη συμφωνία με τις χώρες του Ατλαντικού και μετά θα ασχοληθούν με το TTIP. Για τη χιλή τώρα. Είχαμε μια συνάντηση του Συμβουλίου Σύνδεσης Ένωση Χιλή. Όχι, συγγνώμη, είμαστε σε φάση προετοιμασίας. Θέλουμε να ενημερώσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης στα πλαίσια μιας κοινή ομάδας εργασίας. Θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Μεξικό για την ενημέρωση της αντίστοιχης συμφωνίας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μου. Οπότε, να περάσουμε στο σημείο 4. Η συμμετοχή μας στην ε, κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ στη Γενέβη. Έχετε την έκθεση. συμμετείχαν ε, μια σειρά συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν θέλουμε τώρα να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό, εκτός αν υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν βλέπω. Οπότε παρακαλώ αναφερθείτε στην έκθεση. Αυτό που θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε, ίσως, είναι ότι αυτή η φάση απόλυτης κρίσης ε, του ΠΟΕ φαίνεται ότι, φαίνεται ότι έχει περάσει. Πολλές αντιπροσωπείες μοιάζουν πιο διατεθειμένες να εργαστούν, ε, να δεσμευτούν για συμμετοχή. Αυτό είναι καλό μήνυμα και νομίζω ότι η υπουργική διάσκεψη που θα γίνει το Δεκέμβριο στην Κένια μπορεί να βελτιώσει ακόμη την κατάσταση, άρα η διάσκεψη στη Γενέβη μπορεί να ήταν ένα καλό σημείο έναρξης αυτής της διαδικασίας και να περάσω τώρα στο σημείο 5. Έχουμε εδώ την έκθεση για την επίσκεψή μας στο Βιετνάμ. 6 με 10 Απριλίου και εκεί στείλαμε πολύ άριθμη αντιπροσωπεία. Εγώ είχα την ε, τιμή να ηγηθώ αυτής της αντιπροσωπείας. Συνολικά νομίζω ότι πήγε πολύ καλά, είχαμε πολύ καλές συζητήσεις με εκπροσώπους της κυβέρνησης. Συναντηθήκαμε και με τον Πρωθυπουργό αξιοσημείωτο είναι ότι αναγνώρισε ο Πρωθυπουργό ότι θέλει και δεσμεύεται και είναι προτεραιότητά του η Συμφωνία Ένωσης ε, Βιετνάμ. Ξέρετε ότι το Βιετνάμ διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ και 11 άλλες χώρες στα πλαίσια της Συμφωνίας για τον Ειρηνικό και ο Πρωθυπουργό μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν προβλήματα και μας ε, διαβεβαίωσε ότι η Συμφωνία Ένωσης Βιετνάμ αποτελεί για αυτόν απόλυτη προτεραιότητα. Είχαμε και άλλες συζητήσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα και τους ε, αρμοδίους για οικονομικά θέματα με το Κοινοβούλιο Ξέρετε βεβαίως ότι μια χώρα όπως το Βιετνάμ έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και κατόπιν πήγαμε στην ε, πόλη Χοτσιμίνγκ που είναι το οικονομικό κέντρο του Βιετνάμ πήγαμε σε, μια, σε ένα εργοστάσιο κλωστεφαντουργικών και ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων και συζητήσαμε τις συνθήκες εργασίας. Νομίζω ήταν πολύ επιτυχημένη λοιπόν η επίσκεψή μας. Αυτό βοήθησε σίγουρα την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ίσως λοιπόν τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε ακόμη κάποια ζητήματα που εκκρεμούν, ασάφιες, αλλά με βάση την ισχυρή δέσμευση των ε, συνομιλητών μας είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις και ιδιαίτερα η ομάδα επίβλεψής μας, εποπτείας, πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθεί, να συνοδεύει και να ενθαρρύνει τις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τα ευαίσθητα σημεία όπως κλώστο υφαντουργικά, δασμοί, δικαιώματα εργαζομένων και η επικύρωση των οκτώ κεντρικών προδιαγραφών για εργασιακά του, Παγκοσμίου, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Βεβαίως και ο εισηγητής ε, συμμετείχε και δημιούργησε πολύ συγκεκριμένη εικόνα και θα θέλει οπωσδήποτε να ε, μας πει και αυτό στην άποψή του και να του δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να επιβεβαιώσω όλα όσα είπατε ήδη. Ίσως αξίζει να τονίσουμε ότι η χρονική στιγμή της επίσκεψής μας ήταν ε, ιδιαίτερα κατάλληλη. Πριν την επίσκεψή μας ε, είχαμε ψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου στο Βιετνάμ και συνέπεσε η επίσκεψή μας με την επίσκεψη του Ρώσου Πρωθυπουργού ο οποίος ήταν εκεί μία μέρα πριν από εμάς. Αυτό μας δείχνει ότι το Βιετνάμ ε, είναι τώρα στο προσκήνιο πολλών διεθνών δυνάμεων, δίνεται η προσοχή από πολλές διεθνείς δυνάμεις και φυσικά το Βιετνάμ επικεντρώνεται όχι μόνο στην εμπορική γραμμή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη συνεργασία με την Ευρωσιατική Ένωση και στην γραμμή με τον Ειρηνικό. Πρέπει να τονίσουμε ότι μετά τη Σιγκαπούρη το Βιετνάμ είναι η δεύτερη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας με την οποία προσπαθούμε να ολοκληρωθεί η FTA, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Η αντιπροσωπεία μας έχει τονίσει πολλάκις ότι προτιμούμε ε, να έχουμε ποιότητα παρά ποσότητα ή ταχύτητα και βεβαίως θα είμαστε ικανοποιημένοι αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις εντός ε, του πρώτου εξαμήνου του 2015. Αλλά φυσικά όπως σας είπα υπερισχύει η ποιότητα. Και αν δεν ε, τα καταφέρουμε στο πρώτο εξάμεινο του 2015 θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις ακόμη και την, μετά από αυτή την ε, πιθανή προθεσμία. Συζητήσαμε με βαθμό αξιωματούχου από το Κοινοβούλιο, από την κυβέρνηση, από τον ε, κλάδο της μεταποίησης και της βιομηχανίας, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επίσης, ε, σχεδόν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες ήταν εκεί, το ΕΛ και οι σοσιαλιστές, το ECR, οι φιλελεύθεροι. Δεν ξέρω αν είχαμε πρασίνους και από την ΚΟΕ, δεν νομίζω αλλά νομίζω ότι όλοι είχαν την ε, δυνατότητα να γνωρίσουν την πραγματικότητα του σημερινού Βιετνάμ και μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα οριστικοποιηθούν σύντομα και θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή των όσων έχουμε ήδη διαπραγματευτεί. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάντια. Και τώρα θα δώσω το λόγο ο Ντίβιτ Μάρτιν. Πολύ σύντομα. Καταρχήν σας ευχαριστούμε για την πλήρη ενημέρωση. Σύμφωνα με όσα είπατε, νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η επίσκεψη, αλλά θέλω να αναφέρω κάποια σημεία. Καταρχήν, να αναφερθώ στο τελευταίο σημείο που είπε ο κ. Ζάντια εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι το Βιετνάμ θέλει να συνάψει μια τέτοια συμφωνία μαζί μα και την ικανότητα του να διαπραγματευτεί μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, αλλά έχω σοβαρέ αμφιβολίες για την εφαρμογή, αν μπορεί να εφαρμόσει όσα συμφωνήσαμε. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πέρα από τις διαπραγματεύσεις και την υπογραφή της συμφωνίας σε αυτήν την Επιτροπή, αλλά να δούμε το θέμα της εφαρμογής. Νομίζω ότι με το Βιετνάμ αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με το οικονομικό καθεστώς αγοράς. Όλοι εμείς εδώ συνεχίσαμε να λέμε ότι δεν υπάρχει άμεσο σύνδεσμος μεταξύ της σύναψης μιας FTA και του να αποκτήσει οικονομικό καθεστώς αγοράς η χώρα. Όμως από τη Σκοπιά ε, των ε, Βιετναμέζων ε, μας είπαν όλοι πώς μπορείς να υπογράψεις μια τέτοια συμφωνία μαζί μας χωρίς να μας δώσετε αυτό το καθεστώς αγοράς. Κοιτάξτε, αυτοί πρέπει να σεβαστούν τα κριτήρια ανεξάρτητα από την υπογραφή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει η κυρία Σάπνες. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η επίσκεψη αυτή. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία και την Προεδρία. Ήταν ιδιαίτερα καρποφόρες ε, αυτές οι συναντήσεις. Συμφωνώ με όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Θέλω να προσθέσω τρία σημεία. Καταρχήν όσον αφορά το περιεχόμενο θα πρέπει εμείς να επαγρυπνούμε για το θέμα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπάρχει μια θέση εισαγωγής διακρίσεων απέναντι στην ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία. Μας λένε να καταργήσουμε τους δεσμούς, ενώ το 2018 όλοι οι δεσμοί θα καταργηθούν για το οχήματα που έρχονται από την Νοτιοανατολική Ασία. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα πρέπει να το δεκτούν αυτό. Το δεύτερο θέμα που θα έτω επιτάπητος είναι το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Όλοι το είπαμε με μια φωνή ε, και αν μιλήσουμε πριν το σχάρι για τα ε, κρασιά και ε, για άλλα προϊόντα υπάρχει ένα θέμα προστασίας εδώ που δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα και σχετίζεται και με το θέμα των δικαιωμάτων πνευματικής διοκτησίας. Τρίτον, για τα κλωστοφαντουργικά. Πρέπει να ξέρουμε εμεί οι Ευρωπαίοι ότι τα κλωστοφαντουργικά που θα έρθουν από το Βιετνάμ αν υπογράψουν συμφωνία σε 70% ε, θα έχουν φτιαχτεί στην Κίνα και επομένως ε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις συνέπειες για την ευρωπαϊκή κλωστοφαντουργία και δύο επιπρόσθετες. Μία για το καθεστώ της οικονομίας της αγοράς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχει ε, αυτόματος χαρακτήρας, δηλαδή επειδή θα υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα κτίσουν και αυτό το καθεστώς, θα πρέπει να πληρούνται και άλλες προϋποθέσεις που θεωρώ ότι δεν πληρούνται αυτή τη στιγμή και Κάτι ακόμα, αυτό μα παραπέμπει στη Ατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων σε σχέση με την επίλυση διαφορών μεταξύ κράτου επενδυτή και για τα δικαστήρια. Θα το δούμε αυτό και για άλλε χώρε και άλλε συμφωνίε Η θέση που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη, ίσω και δικαίω αρνούμενη την ε, ιδέα ε, αυτών των ιδιωτικών δικαστηρίων. Ε, κοιτάξτε, εκεί στο Βιετνάμ οι πολιτικοί μα είπαν ε, δεν θέλουμε επίλυση διαφορών μεταξύ του επενδυτή, η δικαιοσύνη θα ρυθμίσει αυτές τις διαφορές. Βέβαια, ε, οι Ευρωπαίοι φυσικά ιδιώτε δεν έχουν την ίδια θέση, δεν θα ρυθμιστεί το θέμα, απλά να το, το, λέμε. Απλώς, ε, ε, το τι θα αποφασίσουμε επί της TTIP θα έχει φυσικά και συνέπειες για άλλες χώρες. Ναι, είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς. Um, um, um We had Ευχαριστώ. Δεν είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην αντιπροσωπεία, όπως και άλλες μικρές ομάδες. Άκουσα όμως πολύ προσεκτικά τα είπατε και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη στο Βιετνάμ. Θέλω να θέσω τρία θέματα. Για να κάνουμε πιο ακριβή τη συζήτηση. Καταρχήν, θα με ενδιαφέρε να μας ε, πείτε ε, τι συνεισφέρει η επίσκεψη στο κεφάλαιο περί ε, που πρέπει να συμπεριληφθεί στην Σύμφωνη Ελευθερών Συνεργών. Γιατί αν μιλήσουμε για το κεφάλαιο περί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Και ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής μας είπε ότι δεν έχει γίνει συγκεκριμένη μελέτη αντικτύπου για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, κάτι που πρέπει να γίνει. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, γιατί δεν έχει γίνει αυτή η μελέτη αντικτύπου εγκαίρως και προβλέπετε το συντομότερο να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή. Δεύτερη ερώτηση για το ISDS επίλυση διαφορών επενδυτή κράτου, ε, συμφωνώ με την κυρία Σάρνε. Λέμε ότι δεν χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο. Τι προβλέπετε λοιπόν, ε, τι συζητάνε οι δύο πλευρές ε, για τη συμφωνία ελεύθερων Συναλλόγων που θα πρέπει να συναυθεί μεταξύ Βιετνάμ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι προβλέπετε αν θα είχαμε τέτοιες διευθετήσεις. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Είχατε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με την κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα, τι περιμένουν και ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η δημόσια συζήτηση στο Βιετνάμ για το θέμα αυτό, έτσι ώστε όταν ε, συζητάμε και διαπραγματευόμαστε για άλλε συμφωνίε, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται. Πολλέ φορέ ε, η κοινωνία των πολιτών δεν γνωρίζει επαρκώ ε, το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και πώ έχει η κατάσταση. Σα ευχαριστώ. Κύριο Βίνκλερ. Ευχαριστώ. Μας κάνατε μια πλήρη παρουσίαση της επίσκεψης της αντιπροσωπείας ε, πολύ σημαντικά. Εγώ θέλω να κάνω κάποια σχόλια πιο συγκεκριμένα. Το θέμα των ίσων κανόνων του level playing field. Αν υπάρχει ή αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο, γιατί αυτή τη στιγμή το καθεστώς των κρατικών εταιριών είναι μια ιδιαιτερότητα της ε, οικονομίας του Βιετνάμ και φυσικά είναι δύσκολο να μιλήσουμε για ε, ίσους κανόνες. Ε, είχαμε μία συνάντηση με τον Περικό στο Βιετνάμ και φυσικά οι απόψεις ε, ότι υπάρχουν εκεί οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στο Βιετνάμ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα να σας πω ότι επισκεφτήκαμε και ένα εργοστάσιο κλωστό υφαντουργίας και θέλω να πω στους συναδέλφους ότι το εισόδημα ενός εργαζόμενου σε ένα εργαστήριο κλωτεφαντουργίας, όχι μόνο σε αυτό που επισκεφτήκαμε, αλλά στην ευρύτερη περιοχή είναι 95% σχεδόν ίσο με το εισόδημα ε, με ενός αντίστοιχου εργάτη, αντίστοιχο εργοστάσιο στη Ρουμανία που είναι κράτος μέλος. Πρόκειται λοιπόν για μια παγκόσμια βιομηχανία, παγκόσμιο κλάδο, αλλά για να δείτε τι συμβαίνει. Τώρα, για την προστασία των επενδυτών, των επενδύσεων. Εγώ εδώ θυαροποθείω από την κυρία γιατί νομίζω ότι να ακούσουμε τι ευρωπαϊκέ εταιρείε στο Βιετνάμ, του επενδυτέ και τι επιχειρήσει, τότε είναι πολύ σαφέ ότι είναι αδύνατο να σκεφτόμαστε ότι το FDS, οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό προστασία των επενδυτών, μπορεί να μην εισαχθεί σε οποιαδήποτε διμερή συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά έχουμε πολύ διαφορετική οικονομία από αυτή της Κίνας, αλλά έχουμε στενές ε, ομοιότητες σε ό,τι αφορά το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. Και τρίτη παρατήρηση, είναι σαφές ότι αν πάει κανείς στο Βιετνάμ θα δει ότι υπάρχει ένας ε, παραλληλισμός ε, μεταξύ της ε, TTIP και της TTIP. Και ίσως το Βιετνάμ θα υπογράψει και την TTP και μεταξύ των 12 κρατών που θα γράψει συμφωνία αυτή μάλλον θα είναι αυτό που θα κερδίσει περισσότερο προς την οικονομική ανάπτυξη. Είναι αυτή λοιπόν μια πραγματικότητα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι ε, έχουμε ουσιαστικά μια προώθηση ε, των διατλαντικών και διερηνικών σχέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Να σας δώσω μερικές ε, συμπληρωματικές για τα θέματα που τέθηκαν. Για την προστασία των επενδύσεων. Όντως, υπήρξε πολύ ενδιαφέρον να διασφαλιστεί η προστασία των επενδύσεων. Αλλά το πώς ακριβώς ε, πρέπει να συζητηθεί. Και σήμερα το απόγευμα φυσικά θα το συζητήσουμε με την Επίτροπο. Και πέρα από αυτό το θέμα, οι επιχειρήσεις, αλλά και άλλοι στο Βιετνάμ, έθεσα το θέμα, αυτό που θα έλεγα άτυπες πληρωμές, δηλαδή πληρωμές που γίνονται έξω από επίσημες δομές. Κάποιος που θέλει να λάβει κάποιες τέτοιες άτυπες χρηματοδοτήσεις. Αυτό λοιπόν θεωρείται από όλους αυτούς σημαντικό πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανόνες για τις επενδύσεις. Είναι θέμα διαφθοράς. Η διαφθορά πρέπει να αντιμετωπιστεί αλλιώς αλλά φαίνεται ότι είναι ένα από τα, μεγαλύτερα, από τα μεγαλύτερα προβλήματα, πέρα από, κάποιες, ε, από κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια. Ναι, Χέλμουτ, βεβαίως. Ε, συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της, Γενομοσπο... της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, αλλά και με προσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Νομίζω ότι αυτή είναι βασική αρχή όλων των επισκέψεων μας. Θέλουμε να έχουμε την ευρύτερη δυνατή εικόνα Υπάρχει μια ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ομάδα 72. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους τους. Οι οποίοι μας ενημέρωσαν ότι όσον αφορά την ελευθερία συνδικαλιστικών οργανώσεων και την ελευθερία έκφρασης ανέφεραν ορισμένα θέματα. Αλλά θεωρούν ότι συνολικά η εξέλιξη είναι θετική. Στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Νομοσπονδίας Συνδικάτων τέθηκε το θέμα του κεφαλαίου βιωσιμότητας. Φυσικά μία νομοσπονδία υπάρχει μόνο στο Βιετνάμ, μόνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουν καταλάβει ότι υπάρχει ανάγκη για μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει, τουλάχιστον θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει, πληθώρα συνδικάτων. Οπότε γι' αυτό το λόγο η Συνομοσπονδία έστειλε μια επιστολή στην κυβέρνηση όπου ε, του ζητά να επικυρωθούν οι οκτώ βασικές ελευθερίες και η ελευθερία λοιπόν του συνεταιρίζεστε που είναι μεταξύ αυτών. Αυτό είναι σημαντικό βήμα για το κεφάλαιο βιωσιμότητας προσωρινά έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες, αλλά θα συμφωνηθούν όλα, εάν βέβαια συμφωνηθούν ακριβώς όλα. Και το βασικό είναι να, επικυρωθεί η... να επικυρωθούν αυτές οι οκτώ βασικές ελευθερίες. Και μετά σίγουρα και το υποπτικό... η εποπτική μας ομάδα θα ασχοληθεί με την εφαρμογή τους. Αυτό θα είναι το κύριο καθήκον της. Και το τρίτο σημείο, σε τι κατάσταση είναι η οικονομία της αγοράς. μου φάνηκε ενδιαφέρον ότι ο πρόεδρος της ε, Οικονομικής Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος μας παρακάλεσε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει οικονομία της αγοράς. Πριν από 20 χρόνια ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Θα αναφερθούμε και πάλι στο θέμα αυτό, θα το συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή. Το θέμα δηλαδή Και είναι οι για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει καθεστώ οικονομία τη αγορά σε σχέση και με τις αποφάσεις που έχει πάρει και η Κίνα βεβαίως σημαντικά και το Βιετνάμ αυτό που λέει για την συμμετοχή τους στον ΠΟΕ που λέει όπως ξέρετε ένα άρθρο ότι μετά από 15 χρόνια καταργείται κάποια ρήτρα και θεωρείται ότι υπάρχει οικονομία της αγοράς. Αυτό βέβαια πρέπει να το εμβαθύνουμε και πολιτικά και νομικά για να έχουμε σαφήνεια. Πολύ ωραία. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό αν δεν θέλει κανείς άλλος το λόγο. Δεν βλέπω. Και να περάσουμε στο σημείο 6. Δυνατότητες του ειδικού τομέα συμβολή στην ανάπτυξη. Εμείς βεβαίως θα ασχοληθούμε κυρίως με τα εμπορικά θέματα και γνωμοδοτούμε προς την Επιτροπή Ανάπτυξης. Υπάρχει μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο που θα μας απασχολήσουν και να δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στην εισηγητριά μας την κυρία Σάντσεθ Καλδεντέη. τα τελευταία χρόνια Βλέπουμε πως ο ιδιωτικό τομέα διαδραματίζει ένα ξενόμενο ρόλο στον ε, τομέα τη ανάπτυξη. Ε, καταρχήν αυξάνονται εμπορικέ παραχωρήσει και ε, κατά την άλλη έχουμε νέα προγράμματα συνεργασία όπου ο ιδιωτικό τομέα έχει πιο σημαντικό ρόλο όπω το blending και άλλοι μηχανισμοί χρήση ιδιωτικών πόρων ή ΣΔΙΤ. Αυτή η διτ αυτη η ταση στην πολιτική συνεργασία συνδέεται με την διεθνή εμπορική πολιτική και αν θέλουμε πράγματι να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη τη στιγμή της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις αρχές της συνοχής πολιτικών για την ανάπτυξη που έχουμε στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τις διεθνείς δεσμεύσεις για την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε την ετερογένεια του ιδιωτικού τομέα γιατί μιλάμε και για τις μεγάλες πολυεθνικές όπως για μικρές και μεσές επιχειρήσεις και τοπικού συνεταιρισμού. Επομένω, δεν έχει τον ίδιο δυναμικό ιδιωτικό τομέα για να συνεισφέρει στην ανάπτυξη που πρέπει να είναι ο πρώτο στόχο. Είναι σημαντικό η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται το πολιτικό χώρο των αναπτυσσόμενων χωρών για να προωθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να δημιουργήσει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, και επικοινομορφία και να ενισχυθεί η ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών για να ενεργοποιήσουν τους εγχώριους πόρους τους. Αυτό θα γίνει αν καταπολεμήσουν τη φορολογική απάτη και τις παράνομες ροές κεφαλαίων. Πολλές φορές αυτό σχετίζεται με τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, την εμπορία ανθρωπίνων όντων ε, και με τα ναρκωτικά. Επίσης ε, θα πρέπει να παρακολουθούμε τι τιμέ των βασικών προϊόντων ε, και να προωθούμε την επιστημιστική ασφάλεια. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία που μπορούν και να περιορίσουν την πρόσβαση στα φάρμακα, να μην αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Αυτό είναι απαραίτητα στοιχεία για να πετύχουμε μια βιώσιμη εσωτερική ανάπτυξη. Επίση, είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπορική τη πολιτική να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση μέσω ενό δεσμευτικού πλαισίου που να εγγυάται ότι οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει θα είναι υπεύθυνε για τι δράσει του σε τρίτε χώρε σε σχέση με του διεθνεί κανόνε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα των φύλων, αξιοπρεπή εργασία, εργασιακά δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντο, πρόσβαση στα φάρμακα, καθολική δυναμική περίθλιψη, πρόσβαση στα τρόφιμα ασφάλεια των τροφίμων. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μία ε, κοινή φωνή. Θέλουμε να ακουστούμε και στην Επιτροπή Ανάπτυξη και ελπίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στίερ, σκιώδης συγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο Λόλα Σάντσεφ που εισήγαγε αυτό το ζήτημα που είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την Επιτροπή μας αλλά και για την καθέληνα αρμόδια Επιτροπή της Ανάπτυξης. Το θέμα είναι ότι φέτος ολοκληρώνουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιτσιρίδας και τους αντικαθιστούμε με ένα νέο σύνολο των επανομαζόμενων στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο βεβαίως να καταπολεμήσουμε και να εκριζώσουμε την ακραία ένδυα. Γνωρίζουμε τώρα ότι η αναπτυξιακή αρρωγή θα ξεκολουθήσει να παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν επαρκεί. Πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα έχει αναγνωριστεί υπό αυτή την έννοια. Αναγνωρίζουμε ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αναγνωρίσαμε πέρσι με ευρία πλειοψηφία ψηφίσαμε ένα ψήφισμα για αυτό το πλαίσιο και αναγνωρίσαμε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικό τομέας. Και βεβαίω σε αυτό το πλαίσιο και το θετικό ρόλο που μπορεί το εμπόριο να διαδραματίσει στην επίτευξη των ε, στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Πάνω 50% των θέσεων απασχόληση παρέχει ο ιδιωτικό τομέα στι ευρωπαϊκέ χώρε. Πρέπει αυτό να το επισημαίνουμε. Και συμφωνώ με τον εισηγήτρια ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές του ιδιωτικού τομέα. Καλό είναι να επικεντρωθούμε στην υποστήριξη των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι επιχειρήσεις γιατί δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και ε, στηρίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα, για άλλε συγκεκριμένε διατυπώσει ε, στο πρώτο προσχέδιο τη ε, εισηγήτρια υπάρχουν κάποια ζητήματα που για το ΕΛΚ αποτελούν κόκκινε γραμμέ, ό,τι αφορά για παράδειγμα την αναθεώρηση των υφιστάμενων συμφωνιών εμπορίου ή τη διατήρηση ισχυρών ε, δασμών εισαγωγικών. Θεωρούμε ότι για την Επιτροπή ΕΝΤΑ χρειάζεται μία διατύπωση που να επικεντρώνεται περισσότερο στις θετικές διαστάσεις ε, των ζητημάτων. Και άλλα σημαντικά θέματα έχουν αναφερθεί, με τα οποία συμφωνούμε, τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και ευθύνη του ιδιωτικού τομέα η λογοδοσία δηλαδή του ιδιωτικού τομέα. Το λεγόμενο blending με την αξιοποίηση διαφορετικών μέσων σίγουρα δεν μπορεί να βελτιωθεί, όμως εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην ε, αναφέρουμε διατυπώσεις που να υπονοούν ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η πρακτική, αλλά να βρούμε τρόπου και λύσεις για να βελτιωθεί η πρακτική. Συμφωνώ επίσης ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε προτεραιότητε, τις επενδύσεις στις πολύ μικρές, μικρές και μισές επιχειρήσεις, γιατί είναι κρίσιμη σημασία και το επαναλαμβάνω και συμφωνώ με τα όσα ανέφερε η συγγήτρια για την προώθηση της ε, χρηστής διαχείρισης και διακυβέρνησης και τη συνεργασία που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ε, άλλες χώρες εταίρους για την οικοδόμηση ανεξάρτητων ε, δικαστικών και δικαιωτικών αρχών. Γιατί θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ευνοϊκό κλίμα για τον ιδιωτικό τομέα για να αναπτυχθεί και με αυτή την έννοια να και για την ευρύτερη ανάπτυξη της χώρας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, καλύτερη και πιο υπεύθυνη διακυβέρνηση. Θα μείνω εδώ. Ήθελα μόνο να τονίσω αυτό το στοιχείο από πλευράς ΕΛΚ ότι το εμπόριο στη θέση μας την οποία θα υποβάλουμε μέσω της Επιτροπής θα πρέπει να ε, επισημάνουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα μας διευκολύνει ε, να επιτύχουμε και τους ε, στόχους μας στους ε, στην Σύνοδο Κορυφής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγητρία για το έργο της. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό κείμενο ιδιαίτερα πλήρες. Και πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε κοινά σημεία και κατόπιν ο καθένας ε, να συνεισφέρει αυτά που θεωρεί πιο σημαντικά για να μπορούμε να καταλήξουμε σε ευρία συνένεση. Εγώ συμφωνώ με όσα λέει η συγγήτρια, σε σχέση ότι μια μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο κύριους άξονες. Καταρχήν, μια καλύτερη ρύθμιση με ρυθμιστικούς δεσμευτικούς στόχους σε σχέση με το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στα σχέδια συνεργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και δεύτερον το να ε, έχουμε να τηρούμε την αρχή της πολιτικής συνοχής. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναλάβει η Ευρώπη και πάλι ηγετική θέση και πολιτική θέση στην αναπτυξία και συνεργασία και εγώ νομίζω ότι σε ένα πλαίσιο ε, δημοσιονομικών περιορισμών ε, οπότε δεν εφαρμόζονται πολιτικές αναπτυξιακές είναι πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε τους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους με μια στρατηγική σημασία που θα χρησιμεύσει για να βοηθήσει την ανάπτυξη στις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, και φυσικά και τις δικές μας επιχειρήσεις να είναι πιο αποτελεσματικές. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερη ρύθμιση. Επομένως θέλουμε ένα σαφέτερο ορισμό για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη συμμετοχή αναπτυξιακά έργα, των κριτηρίων και των μορφών συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Και θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποιους στόχους που θα είναι αηφόροι όσο αφορά την εκτέλεση των σχεδίων που θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα είναι απολύτως διαφανείς και θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Έχοντας ε, αυτά ως κοινά στοιχεία, εγώ θέλω να τονίσω κάποια στοιχεία ε, που νομίζω ότι θα έπρεπε να παρουσιαστούν περισσότερο ή που δεν έχουν αναφερθεί παρκώς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια αναφορά στο είδος της ανάπτυξης που θέλουμε, ε, τι θέλουμε να προωθήσουμε στις τρίτες χώρες. Ε, μια ανάπτυξη που θα τους περιλαμβάνει όλους. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες εμπορίου και επενδυτικές συμφωνίες δεν θα διακινδυνεύουν την ε, πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος από την πλευρά δημοσιοτήτου με εκπαίδευση, υγεία, νερό, ενέργεια. Τρίτον, εμείς πιστεύουμε ότι θα ήταν σημαντικό να υπήρχε μια, ένα μητρό επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναπτύσσουν ε, αναπτυξιακά έργα, έργα αναπτυξιακή συνεργασία, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για το πώ υλοποιούνται αυτά τα έργα, να υπάρχει εχνηλασιμότητα και προκειμένου οι καταναλωτέ να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσει κατάλληλε σε σχέση με το τι καταναλώνουν, ανάλογα με το πώ παρέχονται οι υπηρεσίε αυτέ. Επίσης μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα να μιλάμε και για τη σημασία που έχουν τα δικαιώματα των γυναικών και για την ισότητα των δύο φύλων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ακριβώς οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι χώρες όπου οι γυναίκες υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες κάποιων άδικων και βίαιων δομών. Πρέπει λοιπόν να συνεισφέρουμε με τις αναπτυξιακές μας πολιτικές, στο να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα των δύο φύλων και να φτάσουμε και στην πλήρη ισότητα. Επίσης, δεν συμφωνώ απόλυτα με, τη συνάδελφο, με τον συνάδελφο από το ΕΛΚ σε σχέση με το να μην αναφερθούμε στην αναθεώρηση των σημερινών συμφωνιών. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια αναθεώρηση, δηλαδή να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πώς με τις αναπτυξιακές ε, πολιτικές ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ε, της ζωής των ανθρώπων. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό και θα ήταν σκόπιμο να αναλυθούν οι συνθήκες αυτές. Και τέλος, νομίζω ότι είναι σημαντικό να επιμένουμε στην κοινωνική εταιρική ευθύνη. Και ακριβώ η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και η συνεργασία με το δημόσιο τομέα να βοηθά την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για αναπτυξιακά σχέδια, θα πρέπει να επιλέξουμε επιχειρήσει που να είναι ικανέ, να είναι αποτελεσματικέ από την πρώτη στιγμή για να βοηθήσουν ε, να αναπτυχθεί και ο επιχειρηματικός ιστός, αλλά να αναπτυχθούν και όσοι το χρειάζονται περισσότερο. Γιατί θέλουμε να μπορούν να δημιουργήσουν οι χώρες αυτές ε, τις ε, δικές τους συνέργειες ανάπτυξης. Επιμένω, έχουμε μια καλή βάση επί της οποίας μπορούμε να βρούμε συμφωνία και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σκόπιμο και χρήσιμο να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία ζητώντας από την Κομισιόν αυτά που θέτουμε. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της ε, επίσκεψης ε, στο Βιετνάμ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το ότι χρειάζεται να έχουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, συμφωνώ και εγώ προσωπικά αλλά και η ομάδα μου, νέους και τρόπους εξέτασης της αναπτυξιακής πολιτικής αν Και πώς μπορούμε να κάνουμε τη μετάβαση από τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά μέσα, όπως είναι η οικονομική στήριξη, προς ε, νέα εργαλεία, προς ε, το εμπόριο και τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξή τους. Έχω τις εξής παρατηρήσεις. Κάποιες από αυτές ε, συνάδουν με το πνεύμα της έκθεσης, κάποιες άλλες παρατηρήσεις όχι. Πρώτον, είμαστε Επιτροπή Εμπορίου. Θα πρέπει να επισημάνουμε το ρόλο του ιδιωτικού τομέα και του εμπορίου και της εξωτερικής πολιτικής ως ε, νέου τρόπου για την επίτευξη οικονομικής επιτυχίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Να τους δείξουμε ότι μπορεί έτσι να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός θέσεων απασχόλησης ε, και να αποτελεί αυτό σημαντική πηγή εισοδήματος για τον ε, τοπιο πληθυσμό. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να το τονίσουμε. Δεύτερον, για τους εισαγωγικούς δασμούς, νομίζω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε συζητήσει κατά τη διάρκεια πολλών διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, κατανοούμε και εν μέρη συμφωνούμε ότι οι αναδεσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εισαγάγουν κάποιους ε, εισαγωγικούς ε, δασμούς για να διευκολύνουν την ανάπτυξη της τοπικής τους βιομηχανίας. Από την άλλη όμως, αυτοί οι δασμοί θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι, περιορισμένοι χρονικά και να αφορούν πολύ συγκεκριμένα τις ε, πραγματικά λιγότερο αναπτυγμένες χώρε. Η γενικότερα μεγαλύτερη δασμή ίσως είναι αντιπαραγωγική, θα πρέπει να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Τρίτον, υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Aid for Trade. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικός πάροχος. Και θα πρέπει να αναφέρουμε κάτι για αυτό το στοιχείο στο κείμενο, γιατί είναι μια πολύ σημαντική ε, πρωτοβουλία όπου ενθαρρύνουμε τις ε, σχέσεις business to business μεταξύ επιχειρήσεων. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και τέλος, για την ε, κοινωνική εταιρική ευθύνη. Βεβαίως όλοι συμφωνούν ότι ιδίω οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να λογοδοτούν. Από την άλλη, έχω κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η εισαγωγή δεσμευτικών μέτρων στο εγγραφό μας και αν θα έχουμε έτσι τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, πιστεύω, να καλέσουμε τις επιχειρήσεις να είναι πιο υπεύθυνε, ούτως ώστε ταυτόχρονα μην υπάρχει μεγαλύτερο διοικητικό ή οικονομικό άκτος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν είναι πάντα αυτή η κατάλληλη λύση. Έχουμε προετοιμάσει κάποιες ε, τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ντεσάντας. Ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση είναι επίκαιρη και θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα του ιδιωτικού τομέα και της ανάπτυξης Αρχικά γιατί οι δημόσιες επιχορηγήσεις είναι απαραίτητες, αλλά δεν πρόκειται να αυξηθεί. Θα μειωθεί δεδομένων και των δημοσιονομικών περιορισμών που γνωρίζουμε όλοι. Και αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τους ε, στόχους τη τις παρότι είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε γιατί δεν επιτεύχθηκαν αυτοί οι ε, στόχοι. Πρέπει να το δούμε αυτό πριν περάσουμε στην ε, θέση στόχων για το μέλλον πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό. Θεωρώ ότι ίσω θα μπορούσαμε να εξετάσουμε μια μορφή, διαφορετική μορφή συμπαραγωγή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και αναπτυσσόμενων χωρών και επί τη ουσία δεν είμαι σίγουρη ότι όλη η βοήθεια που δίνουμε, η αναπτυξιακή βοήθεια, όλοι οι δημόσιοι πόροι που δόθηκαν τι τελευταίε δεκαετίε, απέφεραν καρπούς πραγματικά. Πρέπει λοιπόν πράγματι να στηρίξουμε τι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε εντοπίσει, υποδομές, μεταφορικές υποδομές, επενδύσεις, θυματοδότηση, βιώσιμη διαχείριση των ε, φυσικών πόρων και θα πρέπει να υπάρξει και εξέταση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων στι αναπτυσσόμενε χώρε. Μετά, δεν το λέω προκλητικά, αλλά για να το εξετάσουμε. Εδώ και χρόνια χρηματοδοτούμε με δημόσιου πόρου κάποια ε, προγράμματα σε τέτοιε αναπτυσσόμενε χώρε. Για παράδειγμα, στην Κίνα, που χρηματοδοτεί τέτοια προγράμματα, για παράδειγμα, για την οικοδόμηση ενό νοσοκομείου. Πάντα γίνεται με ένα επισυμβαλλόμενο μέρο. για παράδειγμα, το χρηματοδοτεί και μετά ζητάει την ανάπτυξη ενός ε, λιμένα ή ε, μεταφορικού δικτύου. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε μια νέα μορφή εταιρική σχέση που να είναι αμοιβαία επωφελή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Ευχαριστώ. κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή Συμφωνούμε πιστεύω οι περισσότεροι σε μεγάλο βαθμό με την έκθεση. Ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να παίξει ρόλο στην ανάπτυξη. Αλλά να μην υπερτιμούμε το ρόλο του. Δεν είναι πανάκια. Όπως ε, έχουν πει ορισμένοι. Μπορεί να συμβάλλει μόνο εφόσον υπακούει σε σαφείς κανόνες και υπάρχει και εποπτεία. ιδίως όσον αφορά τη φορολόγηση. Η φοροδιαφυγή είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει τους φόρους του. Γιατί μόνο ένα κράτος που έχει πόρους μπορεί να αναπτυχθεί. Πολύ συχνά τι έχω δει σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ευρωπαϊκές εταιρείες που στην Ένωση έχουν καλή συμπεριφορά, είναι καλοί εργοδότες κτλ. Ε, προστατεύουν το περιβάλλον και όταν βγουν από την Ένωση συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι δικές μας εταιρείες ε, τηρούν τα βασικά καθήκοντά τους, για παράδειγμα όσον αφορά τους εργαζόμενους τους και το περιβάλλον. Παντού. Και εμείς ως νομοθέτες έχουμε το ρόλο μας. Βέβαια δεν μπορούμε να επιβάλλουμε νομοθεσία στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά μπορούμε μέσω εμπορικών συμφωνιών, μέσω των κεφαλαίων για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω των επενδύσεων που μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς, ή τη βοήθεια και τις επενδύσεις που μπορούμε να τους δώσουμε, να διασφαλίσουμε να υπάρχει υποχρεωτική υποβολή έκθεση χώρα ανά χώρα για όλες τις εταιρείες, διαφάνεια, οι φορολογικές αποφάσεις, συμμόρφωση με το εθνικό δίκαιο, όλα αυτά πολύ σημαντικά και θα πρέπει να υπάρχουν σημεία επαφή όσα για να αποστέλλονται τα παράπονα. Πολλά πρέπει να κάνουμε και να βελτιώσουμε και τους μηχανισμούς εποπτείας για το σεβασμό των συμβάσεων του Παγκοσμίου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασία. Βέβαια το ISDS το συζητάμε πολύ. Παίζει όμως ρόλο και στις αναπτυσσόμενες χώρες γιατί μόνο εάν υπάρχουν σωστές συνθήκες μπορούν να αναπτύξουν την κοινωνική τους νομοθεσία, την προστασία των καταναλωτών. Να μην το ξεχνάμε όταν συζητάμε το ISDS. Θα υποβάλουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά συνολικά συμφωνούμε με τη βασική κατεύθυνση και ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντική έκθεση αυτή Χαίρομαι και για τον ε, γύρο της ΔΟΑ. Νομίζω ότι ο αναπτυξιακός γύρος ε, βοήθεια για το εμπόριο έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία πέρα από τη διευκόλυνση του εμπορίου αυτοί οι τομείς είναι οι τομείς που μπορούν να βοηθήσουν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τονίζουμε πάντα ότι σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι στην Γενέβη και ελπίζουμε μέχρι το Δεκέμβριο που θα έχουμε τον, ε, τη συνάντηση του ΠΟΕ να έχουμε σημαντικές πολυμερείς επιτυχίες και πρόοδους και επίσης η κατάργηση των ε, δασμών χρειάζεται λειτουργικές εφορίες για να μην γίνονται καταχρήσεις και για να μην ε, εκμεταλλεύονται κάποιοι την κατάσταση. Ούτως ή άλλως είναι βασική προϋπόθεση η επαρκής λειτουργία των φορολογικών αρχών για την μόνιμη ανάπτυξη των χωρών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο και στην Κομισιόν, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος, είναι παρόν για να την εκπροσωπήσει. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι υπεύθυνο στην ΔΕΒΚΟ, τμήματάρχη για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη γνωμοδότηση και τις απόψεις που αναφέρθηκαν για τον αυξανόμενο ρόλο του ειδικού τομέα για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πέρυσι εγκρίναμε μία ανακοίνωση που αναφέρει τις ε, σαφείς αρχές και κριτήρια για τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη και πώς θα πρέπει να είμαστε σε επαφή με τον ιδιωτικό τομέα για να έχει αναπτυξιακούς στόχους. Και αυτές οι αρχές και τα κριτήρια συμπληρώνουν τις αρχές της ε, διεθνούς αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας και τονίζω ότι το άρθρο 208 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως την πολιτική μας και επίσης, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στη συζήτηση που γίνονται τώρα διεθνώς για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και για την κατάσταση μετά το 2015. Ο ρόλος λοιπόν αυτός είναι σημαντικός. Για τα σχόλια του εισηγητή, συμφωνώ με πολλά σημεία που ανέφερε και νομίζω ότι συμβαδίζουν με την ανακοίνωσή μας Και τονίζω, τονίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολύ διαφορετικοί ε, πολύ διαφορετικές εταιρείες οπότε η διακυβέρνηση και η λήψη υπόψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι στην καρδιά των προγραμμάτων μας. Στη γνωμοδότησή σας αναφέρεται ότι οι πρακτικές μας για να μοχλευτεί η ιδιωτική χρηματοδότηση δεν έχουν καταλήξει ακόμη, δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Οι βασικές αρχές που αναφέρονται στην χρηματοδότηση είναι και στην ανακοίνωση. Όλα αυτά είναι στη βάση της πολιτικής μας, οι πολιτικές συνδυασμού δηλαδή. Καμία από τις αποτιμήσεις και αναθεωρήσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν συνδέουν ε, την ανεπαρκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με την έλλειψη διαφάνειας ή την παραβίαση κάποιας άλλης από τις αρχές. Τώρα για την εμπορική πολιτική. Βεβαίως μπορεί να, να ενισχύσει, να στηρίξει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη. Και φυσικά σε όλες τις συμφωνίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι όλων των συμβαλωμένων και ως Επιτροπή πάντα δεχόμεθα ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να υπερασπιστούν και να προστατεύσουν τους πιο ευαίσθητους τομείς της οικονομίας τους. Τώρα δεν ξέρω εάν ε, η υψηλή εισαγωγική δασμή είναι ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχουν αυτό. Αυτό πρέπει να το δούμε αναπερίπτωση μέσω μελετών επιπτώσεων. τα κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης ε, συστηματικά συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες. Αυξανόμενη λοιπόν η σημασία αυτού του τομέα, χαιρετίζω τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, θα λάβουμε υπόψη τον αυξανόμενο ρόλο του ιδιωτικού τομέα κατά την εφαρμογή των στόχων μας για την περίοδο 30-40 με βάση τις αρχές και τα κριτήρια στα οποία προαναφέρθηκα και τα οποία περιλαμβάνουμε στην ανακοίνωσή μας και βεβαίως σημειώνουμε με πολύ σοβαρότητα τη συζήτηση σήμερα. Επιστρέφουμε στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσει με τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Περιμένω τις τροπολογίες τους για να αρχίσουμε να εργαζόμαστε επί των συνδυασμών για να απαντήσω στον πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί το ελεκτικό συνέδριο ε, αναφέρθηκε στο θέμα του συνδυασμού των μέσων και της διαφάνειας σε μια μελέτη και τον θεσβήτησε. Γι' αυτό το έχουμε συμπεριλάβει στο σχέδιο κειμένου της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας και ελπίζουμε να έχουμε μια ισχυρή άποψη που θα ακουστεί στην Επιτροπή ε, Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Προθεσμία για τις τροπολογίες 8 Μαΐου. 12 το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε στις 28 Μαΐου. Θα έχουμε αρκετό χρόνο μετά, τη συμφωνία, μετά την ψηφοφορία για το TTIP. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στο σημείο αυτά. Ετήσια έκθεση για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και να δώσω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Μπορέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι προκλήσεις που μας ε, τίθενται σήμερα καθεστούν προφανές ότι η αρχή της επικουρικότητας λαμβάνει μια νέα διάσταση και θα πρέπει να είναι στοιχείο ισορροπίας μεταξύ ε, των αρμοδιοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο και την απέτηση των πολιτών να έχουν περισσότερο έλεγχο και επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Η έκθεση 2013 που παρουσιάστηκε από την Κομισιόν ε, δεν ασχολήθηκε με την αρχή της ε, επικουρικότητας στην εμπορική πολιτική, έτσι αυτή να εννοηθεί ότι αυτή είναι αποκλειστική κοινοτική αρμοδιότητα. Εμείς θέλουμε να θέσουμε ακριβώς αυτό το θέμα προτείνοντας τους εξής προβληματισμούς. Καταρχήν, οι προκλήσεις που μας τίθενται σήμερα απαιτούν να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο από το παρελθόν, ε, θέτοντας στο προσκήνιο όλα τα πολιτικά παραδείγματα που διαθέτουμε και μεταξύ αυτών την αρχή της επικουρικότητας. Δεύτερον, η αρχή της επικουρικότητας είναι ένα οριζόντιο στοιχείο σε όλες τις πολιτικές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αποκλείεται από την εμπορική πολιτική και επίσης η μη ισορροπημένη χρήση της στα μέσα δημόσιας διαβούλευσης και μελέτης αντικτύπου από ορισμένες υπηρεσίες της Κομισιόν. Επομένως, αυτό είναι σημαντικό γιατί χωρίς σοβαρή ανάλυση του αντικτύπου και των αποφάσεων που μπορεί να, που μπορεί να υπάρχει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό κινδυνεύει να απομακρύνει ακόμη περισσότερο τους πολίτες από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών ζητούν περισσότερη ενημέρωση και διάλογο με τα θεσμικά όργανα. Αυτή η διάσταση είναι η πρόκληση της επικοινωνικότητας που έχουμε ενώπιόν μας. Επομένω, με αυτό το πνεύμα και τη συνειδητοποίηση, εγώ θέλω να σας παρουσιάσω συντομία κάποιες σκέψεις που έχουμε στην έκθεση για την επικορικότητα του 2013, στεκόμενος ιδιαίτερα σε πέντε σημεία. Το πρώτο σημείο αφορά το ρόλο της ε, ε, επικουρικότητας ε, στις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βάσει των πολλαπλών συμφωνιών που συνάπτει η Ένωση με τρίτες χώρες. Η επικουρικότητα λαμβάνεται υπόψη όταν υπάρχουν διατάξει διεθνών συμφωνιών που έχουν αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο και επομένω, απαιτούν από τα κράτη-μέλη να τοποθετηθούν. Αν και με τη συνθήκη τη Λισαβόνα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε αποκλειστικέ αρμοδιότητε σε θέματα εμπορική πολιτική, παρόλα αυτά υπάρχει ένα χώρος αβεβαιότητας εκεί όπου μια εμπορική συμφωνία προβλέπει διατάξεις που δεν αφορούν αποκλειστικά τις εξωτερικές, τις άμεσες εξωτερικέ επενδύσεις όπως μας έδειξαν πρόσφατες συμφωνίες με τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όπου μπορούν να ανακύψουν κάποιες συγκρούσεις αρμοδιότητας και επομένως εμεί θεωρούμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ιδίως σε ορισμένους κλάδους όπως της ενέργειας. Ε, μια άλλη πτυχή αφορά τις ρήτρες διασφάλισης και τις πιθανές συνέπειες κορικότητας όπως μας δείχνει η συμφωνία με την Νότιο Κορέα. Το δεύτερο θέμα αφορά τη μακροοικονομική βοήθεια. Ε, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην εξωτερική πολιτική. Πολύ συχνά η ιδεολογική συζήτηση μας εμποδίζει να επικεντρωθούμε στις συγκεκριμένε συνέπειες αυτή. Το κριτήριο της επικουρικότητας μας ζητά να αξιολογήσουμε προσεκτικά αν οι προτάσεις μας μπορούν πράγματι να είναι χρήσιμες για τους εταίρους που βοηθούμε. Φυσικά μετά από μια προσεκτική εξάντη ανάλυση και ε, φυσικά με επαρκή έλεγχο του Κοινοβουλίου για τη χρήση των πόρων μπορούμε να αναφέρουμε την αρχή του More for More που υιοθετήθηκε για τη βοήθεια στις χώρες της Μεσογείου κατά τη διάρκεια της αραβικής άραξης που κατόπιν αποδείχθηκε ήταν εντελώ αποτελεσματική. Το τρίτο σημείο αφορά την αναγκαιότητα να ξαναδούμε τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η μελέτη αντικτύπου εξάντε για τις εμπορικές συμφωνίες. Πολλές φορές δυστυχώς συνεχώς έχουμε καταπληκτεί από ε, ιδιαίτερα αισιόδοξε μελέτες αντικτύπου ε, και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στη συζήτηση για το TTIP. Οι διαπραγματεύσει ξεκίνησαν το 2013 για το TTIP. Είναι με σαφές ότι έχει πολύ μεγάλη πολιτική ε, αξία μια τέτοια συμφωνία γιατί συνδέει στρατηγικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Όμως είμαστε σίγουροι ότι είναι χρήσιμη με τη συμφωνία για τις επιχειρήσεις και και τους πολίτες μας. Είμαστε σίγουροι ότι έχει θετικές συνέπειες για όλους εμάς και όχι μόνο για τις λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το θέμα. Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γιατί οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν ε, βάσει εκτιμήσεων που δεν μπορούν ούτε να αποδεικτούν ούτε να αποσυντικοποιηθούν μέσω της μεθόδου ανάλυσης που θέτει η Κομισιόν. Και επομενω στην περίπτωση αυτή περισσότερο από ποτέ η αρχή τη επικορικότητας και της πρόληψης θα πρέπει να είναι στη βάση οποιασδήποτε διαπραγμάτευση της Κομισιόν. Πολλές φορές η αξιολογήσει των περιβαλλοντικών αντικτύπων, κοινωνικών ή κοινωνικών αντικτύπων λείπουν στην αρχή της διαπραγμάτευσης και γίνονται μόνο κατά τη διάρκεια. Έτσι λοιπόν ε, θα έπρεπε στο προκαταρκτικό σχέδιο της διαπραγμάτευσης να γίνεται κάτι τέτοιο για να καταλάβουμε πλήρως ε, τη συνέπεια της ε, συμφωνίας. Μια, ένα άλλο στοιχείο έχει να κάνει με την επίλυση διαφορών κράτους επενδυτή. Εδώ έχουμε σύγκρουση η μεταξύ ε, της ε, κυριότητας ε, των κρατών μελών και της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ πρέπει να αναλυθεί αυτό πλήρως σε σχέση με την τύπη. Το τελευταίο σημείο με το οποίο θέλω να κλείσω αναφέρει πάλι ένα θέμα σημαντικό σε μένα και που βρίσκεται στην καρδιά της επικουρικότητας. Είμαι πεπισμένος ότι ο καθένας από εμά εδώ, σε αυτό το κοινοβούλιο, έχει ε, εκπροσωπώντας ε, άμεσα του ψηφοφόρους ε, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους και όλα τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω όταν ε, μιλάμε για το θέμα της επικουρικότητας πανίως μιλάμε για τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο. Θέλω λοιπόν να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι πολίτες στη διαδικασία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε θέματα εμπορική πολιτική. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση πρόκληση της Οι πολίτες θέλουν περισσότερες πληροφορίες και να εμπλέκονται περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κυρίως όταν υπάρχουν ενδυνάμεις συνέπειες για τα μέσα συμφέροντά τους. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά μέσα για να ενημερώσουμε τους πολίτες και να τους εμπλέξουμε και αυτό το στοιχείο δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Φυσικά δεν αρκεί η δημόσια διαβούλευση που χρησιμοποιείται από την Κομισιόν γιατί δεν εγγυάται μια ισορροπημένη συμμετοχή. Αν οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες ε, θέλουν να είναι όσο δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη, ε, σίγουρα θα είναι πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες συγκεκριμένες και θετικές. Στο φως αυτό το σκέψεων σας προτείνω τον εξή προβληματισμό ξεκινώντας από τη μελέτη αντικτύπου ε, που θα γίνεται με έναν τρόπο που θα σέβεται περισσότερο τις διαδικασίες de facto και de jure, μπορούμε να έχουμε δημόσιες διαβουλεύσεις που θα είναι πραγματικά σημαντικές και θα μας δείχνουν ποια είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα και ουσιαστικά μία ε, δημόσια διαβούλευση για να ισχύει θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα σύστημα της δυτής πλειοψηφία που εφαρμόζεται και στο Συμβούλιο. Έτσι η αρχή που θα εφαρμοστεί για την εμπορική πολιτική μπορεί να καλύπτει αυτό το χώρο δράση που αφήνουν οι συμφωνίες και ε, θα έχουμε μελέτες αντικτύπου που θα λαμβάνουν υπόψη και την τοπική διάσταση και θα έχουμε δημόσιες διαβουλεύσεις που θα είναι πράγματι σημαντικές. Μπορεί να μας φαίνεται δύσκολη αυτή η πρόκληση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα ε, να προβλέπουμε τα μελλοντικά προβλήματα και ότι μια διαχείριση της επικουρικότητας με έναν και αποτελεσματικό τρόπο μπορεί να είναι ένα σημαντικό σημαντικό στοιχείο ε, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της κοινότητάς μας, ε, των κοινότητων μας. Σας ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο τώρα στους κοιόδης. Ο κύριος Χουές. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες σκέψεις για την έκθεση του κυρίου Μπορέλη γενικά συμφωνούμε με τις προτάσεις που παρουσιάζει στην εκθεσή του για το θέμα αυτό. Επίσης συμφωνούμε με την έμφαση που έδωσε και επανέλαβε μόλις για το πρόβλημα της επικουρικότητας. Αυτό το θέμα βέβαια της επικουρικότητας ε, δεν είναι και πολύ σχετικό με την κοινή εμπορική πολιτική. Αυτό δυνάμει τη συνθήκη, ε, γιατί έχουμε αποκλειστική ερμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο βαθμό αυτό πρόκειται για μια πραγματικά κοινοτική πολιτική. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι ε, έχουμε ορισμένα στοιχεία που πρέπει να δούμε. Αναφέρθηκε, παραδείγματος χάρη, μακροοικονομική βοήθεια σε τρίτες χώρες που προβλέπεται από το άρθρο 202 ή και η σύναψη μεικτών συμφωνιών με τρίτες χώρες, όπου οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας λαμβάνουν ε, ένα σημαντικότερο χαρακτήρα και θα πρέπει να γίνονται σεβαστές σε ό,τι αφορά τώρα τα αιτήματα μακροοικονομικής βοήθειας, συμφωνώ με την ιδέα ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια καλύτερη αξιολόγηση αντικτύπου, εξάντε, κυρίω όταν βρισκόμαστε ενώπιον καταστάσεων αναλογικότητας και όταν η οικονομική βοήθεια δεν, ε, πρέπει να δίνεται κατεπηγόντως. Επίσης, ε, θέλω να αναφερθώ στο ότι είναι σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε θεσμική ισορροπία. Φυσικά, σε ό,τι αφορά αυτή την κοινή εμπορική πολιτική, πρέπει να διατηρήσουμε, όπως σας είπα, διοργανική ισορροπία, δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών και κρατών μελών βάσει της δίκης ε, της Ρώμης ε, πρέπει να διατηρήσουμε αυτό που προβλέπονται ως προς ε, την κοινοτική αρμοδιότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εργασία μέχρι τούδε. Πολύ ενδιαφέρουσα. Και σε βαθμό συμφωνώ ιδιαίτερα αυτά που είπατε για τα θέματα που έχουμε με τις μελέτες επιπτώσεων. Δεν είναι αντικειμενικές, είναι υπεραισιόδοξες αυτές οι μελέτες αντικτύπου. Και οι συγκρούσεις για θέματα αρμοδιότητας μεταξύ κρατών μελών και ένωσης. Και εδώ χρειάζεται βελτίωση, ιδιαίτερα για κάποιες συμφωνίες για τις ε, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είμαστε θετικοί. Αλλά θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για να βελτιωθεί η ισορροπία του κειμένου. Αλλά να πω κάτι συνολικά για αυτά που είπατε για την επικουρικότητα. Για μένα η επικουρικότητα σημαίνει ότι τα θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται εκεί που είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται η εμπορική πολιτική της Ένωσης και άμα αν τη συγκρίνω με την εξωτερική πολιτική έχω την εντύπωση ότι λειτουργεί πολύ καλύτερα η εμπορική πολιτική. Είμαστε εμπορικοί υπερδύνομοι. Ενώ είμαστε πολιτικά ανάνος γιατί κάθε κράτος μέλος δεν... κάθε κράτος μέλος συγγνώμη, ε, συμπεριφέρεται διαφορετικά. Εγώ δεν νομίζω λοιπόν ότι εάν κάτι ρυθμίζεται σε επίπεδο κράτους ε, ε, αντιμετωπίζεται καλύτερα, ούτε αν αντιμετωπίζεται σε επίπεδο περιφέρειας, κατά ανάγκη αντιμετωπίζεται καλύτερα. Κοιτάξτε, βεβαίω, ε, μέσω αυτών των συμφωνιών ISDS μπορούν πολλά να κερδίσουν οι δικηγόροι. Αλλά δεν νομίζω ότι η λύση θα ήταν κάθε κράτος μέλος πρέπει να αντιμετωπίζει από μόνο του και διαφορετικά τα θέματα αυτά διαφωνιών, επενδυτών και κράτους. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα καλύτερα. Διαφορετικά από ό,τι ήθελε αρχικά η κυρία Μάνστρομ και θα ακούσουμε τα απόγευμα θα μας πει. Αλλά πρέπει να υπάρχει περισσότερη ισορροπία. Νομίζω σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα στον εμπορικό τομέα είναι λάθος η και χωρισμένη αντιμετώπιση. Εκεί που έχετε δίκιο είναι ότι πρέπει να συμμετέχουν και να ενημερώνονται οι πολίτες. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Αν ε, είμαι κατά του ISDS δεν είμαι μόνο για τους Αυστριακούς που δεν τη θέλουν. Είμαι ε, επίσης εκπροσωπώ και τους πολίτες άλλων χωρών που δεν τη θέλουν. Επ' αυτού του σημείου λοιπόν διαφωνώ, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι η έκθεση είναι αρκετά καλή. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω να λείπουν διάφορες σκιώδεις τώρα. Οπότε είναι ο κύριος Μπούχνα. Α, είναι παρόν. Α, συγγνώμη. Α, δεν με ενημέρωσαν. Αλλά παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης εκ μέρους της ομάδας μας, γι' αυτό παρευρίσκομαι. Ε, ήθελα να προσθέσω δύο λόγια στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Ουσιαστικά κάποιες διευκρινήσεις που νομίζω ότι είναι απαραίτητες. Η έννοια της επικουρικότητας πολύ συχνά πολιτικοποιείται προβολικά. Και ιδίω ό,τι αφορά το εμπόριο υπάρχουν πολλοί τρόποι που οι πολίτε και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να επηρεάσουν του υπουργού όταν εξετάσουν ε, αυτά τα ζητήματα ή παίρνουν αποφάσει στο Συμβούλιο. Και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσωπούμε του πολίτε από όλο το πολιτικό φάσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα μία διευκρίνηση για το τι ακριβώς σημαίνει η αρχή, η αρχή της συναλλογικότητας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε, ότι εργαζόμαστε από κοινού στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική και τι διαπραγματεύσει με τρίτε χώρες, αυτό ε, δημιουργεί όφελο για μα. Κανένα κράτο μέλο δεν μπορεί να πιστέψει ότι ε, αν πήγαινε από μόνο του να κάνει διαπραγματεύσει με τρίτε χώρε θα είχε την ίδια διαπραγματευτική ισχύ. Και μετά υπάρχει μια αναφορά σε κάτι άλλο που δεν το γνωρίζω καλά. Τι εννοείται με τις ε, διμερείς ρήτρες ασφαλείας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Υπάρχει στη συνθήκη της Λισαβόνας, είναι επιπρόσθετα μέτρα που προτείνεται. Δεν κατανοώ τι εννοείται με αυτή τη δικλίδα ασφαλείας και μετά υπάρχει αναφορά στο προσχέδιο στην αρχή ή την αρμοδιότητα λήψη αποφάσεων. Και μετά για τις συζητήσεις αυτές που αρκετά πολιτικές γίνονται, τελικά υπάρχει και νομικό ζήτημα. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή μπορούν να ζητήσουν ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αν υπάρχει αβεβαιότητα ή διαφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε τα νομικά και τα πολιτικά ζητήματα πιο ξεκάθαρα εδώ. Υπήρξαν σχόλια για τις εξολογήσεις αντικτύπου και στο σχέδιο κειμένου. Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να δούμε πού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει από μόνη της τη μελέτη και πού ε, αναθέτει την εκπόνηση μιας μελέτης σε εξωτερικούς ε, φορείς, πανεπιστήμια και το καθεξής. Είναι δύσκολο ότι όλα αυτά τα στοιχεία γίνονται με πολιτικό γνώμονα. Πρέπει να δούμε σε ποιον απευθυνόμαστε εδώ. Και μετά πρέπει να δούμε τι συνέβη στο παρελθόν με τι εμπορικέ συμφωνίε, γιατί η αξιολόγηση της, ε, του αντικτύπου του εμπορίου δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα και πάντα εξαρτάται από πολλαπλού παράγοντε. Ποτέ δεν μπορούμε να τα καλύψουμε αυτά κατά 100% σε οποιαδήποτε μελέτη. Είναι επιστημονικά αδύνατον. Όμω φέρουμε την ε, παρελθοντική μας ε, εμπειρία. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφεληθεί τα μάλα από το διεθνέ εμπόριο. Πρέπει λοιπόν να τα εκτάσουμε και αυτό. Ακόμα δύο σημεία. Αναφορά στην αρχή more for more που ανέφερε. Αναφερθήκε σχετικά. Η εμπορική πολιτική είναι ένα, ένα στοιχείο που αξιοποιείται σε όλο το φάσμα της εμπορικής μας και εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λογοδοσία για τους πόρους, ε, τα μέσα και την χρηματοδοτική βοήθεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε ευρύτερα, δεν είναι μόνο εμπορικό θέμα. Μετά γίνεται αναφορά στην ε, ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχή και σύνδεση και συμπερίληψη των ε, ενδιαφερμένων μερών. Αυτό είναι κάτι το οποίο με βρίσκει σύμφωνη ως αεστόχος. Να δούμε τις προσδοκίες, το ενδιαφέρον. Ε, υπάρχει ανάγκη να υπάρχει σε μεγαλύτερη διαφάνεια, όμως πρέπει να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε αυτό. Αν έχουμε πολύ διαφορετικές προσδοκίες μια ομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τη αφορά το προπολογισμό ή το προσωπικό τη, πρέπει να δούμε και τι είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι εννοεί ο συγγητή. Θέλει να διαθέσει περαιτέρω πόρου για να διαμορφωθεί και αυτή η ικανότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει σκιώδης από την ΚΟΕ. Δεν είναι εδώ σκιώδης μας, αλλά μπορώ να κάνω μια, ένα σύντομο σχόλιο. Αλλά μετά από τους ε, υπόλοιπους σκιώδης. Ο κύριος Βούπνερ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτά που είπε κυρίως για την συμπερίληψη της κοινή γνώμης στα κράτη-μέλη. Και εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Από πλευρά τη ομάδα μου η ιδέα ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα να μπουν στην ε, εμπορική πολιτική είναι μια τολμηρή ιδέα, αλλά θα είμαστε ατεθειμένοι σε έναν βαθμό να συμφωνήσουμε και θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο εργασίας μας ως Επιτροπή Εμπορίου. Όμως από την ε, επιχειρηματολογία της παραγράφου 32 δεν συμφωνώ. Αυτό το είπε και κάπως ο εισηγητής Πρώτα απ' όλα θέλουμε να αποφασίσει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρμοδιότητα που υπάρχει που δόθηκε για τα θέματα αυτά για τις επενδύσεις, δηλαδή τις αρμοδιότητες για τις επενδύσεις που δόθηκε από την ε, ε, συμφωνία συγγνώμη, από τη συνθήκη της ε, Νίκαιας διότι ξέρετε ότι στις ε, συνθήκες μας ε, είναι γενική αρχή η επικουρικότητα η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν ένα θέμα δεν έχει ρυθμιστεί πλήρως από τις συνθήκες. Άρα εδώ μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, αλλά ενδιαφέρον. Στην τέταρτη και πέμπτη παράγραφο και την τελευταία φράση της δεύτερης ε, παραγράφου συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με την ε, επιχειρηματολογία για την αλογικότητα και θα είμαστε, για, ε, είμαστε διατεθειμένοι να υποβάλουμε τροπολογίες. Ε, συμφωνούμε με το κείμενο της έκτης παραγράφου, αν και δεν νομίζουμε ότι με τη στενή έννοια αφορούν, ε, αφορά αυτή η παράγραφος την επικουρικότητα και την αλογικότητα. Ευχαριστώ από την Επιτροπή κύριος Μπόρν. Ο Χέλμουντ θέλει ακόμη το λόγο. Ο Χέλμουντ Σόλτ. Όχι, ήθελα να μιλήσω. Απλώς ήθελα να αφήσω να μιλήσουν πρώτοι οι σκιώδει. Δεν ήθελα λοιπόν να μιλήσω πριν από αυτούς. Σε δύο θέματα λοιπόν θέλω να αναφερθώ. Για αυτά που είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένω. Πρώτον, σωστό είναι ότι η επικουρικότητα είναι αρχή. Αρχή που αναφέρεται στις συνθήκες. Πρέπει λοιπόν κατόπιν να δούμε συγκεκριμένα ποια θέματα εμπορικής πολιτικής είναι ενωσιακή αρμοδιότητα και λόγω της επίπτωσης ε, της ε, εμπορικής πολιτικής στην οικονομική, κοινωνική τα κατάσταση στα κράτη-μέλη θέλουμε να υπάρχει και μια κρατική, εθνική αρμοδιότητα να μπορούν να ελέγξουν τι επιπτώσεις έχει δηλαδή η εμπορική πολιτική. Οπότε συμφωνώ επ' αυτού με πολλές παρατηρήσεις πολλών συναδέλφων. Επίσης θεωρώ ότι επέλεξε ενδιαφέρουσα προσέγγιση ο εισηγητής, αλλά να αναφέρω ένα επιπλέον σημείο. Το αναφέρει η μακροοικονομική βοήθεια. Τη συγκεκριμένη χρήση της διαπιστώσαμε ότι τους τελευταίους μήνες συμφωνήσαμε ότι πρέπει να έχουν κάποια δυνατότητα να επιδράσουν τα κράτη-μέλη, αλλά όχι αναδρομικά. Ξέρουμε ότι έχει επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των χωρών η εμπορική πολιτική, αλλά αντίστροφα θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ίσως θα έπρεπε να το διευκρινίσει κάπως περισσότερο ο εισηγητής. Πού θέλει να αλλάξει η κατάσταση σε σχέση με τις εκπεφρασμένες ε, ρήτρες της συνθήκης. Σε ποια σημεία θεωρεί ότι χρειάζεται τροποποίηση των συνθήκων λόγω της επίπτωσης στην πραγματική κατάσταση οικονομίας θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο αντιμετώπισης εμπορικής πολιτικής. Νομίζω πως είναι σημαντικό σημείο αυτό και θα, θα συμμετάσχουμε στην περαιτέρω εξέταση της έκθεσης. Και τώρα ο κύριος Μπάρν, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Εκ μέρου τη Επιτροπή θα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, του κοιόδη εισηγητέ και τα μέλη για τι παρατηρήσει του σε αυτό το σχέδιο έκθεση. Θα ήθελα να ομοδοποιήσω τι παρατηρήσει, αρχικά γύρω από το ζήτημα τη επικουρικότητα και δεύτερον στο ζήτημα του, της αξιολόγησης αντικτύπου. Όπως είναι γνωστό, η αρχή της επικουρικότητας εγγράφεται στις ε, στη συνθήκη. Η συνθήκη διευκρινίζει πού και με ποιο τρόπο εφαρμόζεται η αρχή, η αρχή της επικουρικότητας. Η εν λόγω έκθεση που αναλύει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει προετοιμαστεί από την Επιτροπή και εξετάζει την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Η έκθεση δηλαδή δεν εξετάζει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να ισχύει η αρχή της επικορικότητας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιδιαιτερότητα της επικορικότητας στο πλαίσιο της ομπρικής πολιτικής. Όπως ε, αρκετά μέλη ανέφεραν, το εμπόριο είναι ζήτημα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή της επικουρικότητας αυτή καθ' αυτή δεν ισχύει Αναφέρθηκε προηγουμένως ε, ένα καλό παράδειγμα αιτιών γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια κοινή πολιτική εάν το ένα κράτος μέλος έχει μια προσέγγιση ότι φορά την απελευθέρωση των δασμών και ένα άλλο κράτος μέλος διαφορετική προσέγγιση. Πρέπει να έχουμε λοιπόν κοινή πολιτική και αυτό ε, απαιτεί το να αποτελέσει θέμα αποκλειστική αρμοδιότητας. Και έτσι η αρχή τη επικουρικότητας δεν ισχύει στο πεδίο αυτή τη αποκλειστική αρμοδιότητας. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή έχει ζητήσει νομοδότηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ε, ισορροπία αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών για να διευκρινιστούν αυτά τα ζητήματα. Κάποια σημεία θα πρέπει να τα επισημάνουμε σε ό,τι αφορά την ε, αλληλεπίδραση μεταξύ εμπορικής, πολιτικής και αρμοδιοτήτων κρατών μελών. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η εμπορική πολιτική παρέχει ένα πλαίσιο θεσπίζει ορισμένου κανόνε που την χάνουν διαπραγμάτευση σε διεθνέ επίπεδο. Και αυτή η αναφορά ε, στην παράγραφο 3 τη έκθεση δεν διακυβεύει τι αρμοδιότητε των κρατών μελών, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τι ε, περιβαλλοντικέ πολιτικέ ή πολιτικέ ε, υγεία ή στο πλαίσιο της επίλυσης διαφορών κράτους επενδυτή δεν διακυβεύεται η δικαιοδοσία του Εθνικού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά το εθνικό δίκαιο. Το ISDS είναι θέμα εφαρμογή διεθνού. δικαίου. Θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τις ε, αξιολογήσεις αντικτύπου. Η έκθεση της Επιτροπής που αποτελεί τη βάση ανάλυσης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων εξετάζει τις αξιολόγησεις αντικτύπου αλλά και το έργο της Επιτροπής για την ανάλυση της επικουρικότητας στο πλαίσιο της αξιολόγησης αντικτύπου. Δεν είναι δηλαδή μια έκθεση για την γενική ε, λειτουργία ε, των αξιολογήσεων αντικτύπου και αν θα πρέπει να βελτιωθούν ή όχι. Δύο παρατηρήσεις πιο συγκεκριμένα για το ζήτημα των αξιολογήσεων αντικτύπου. Πρώτον, να είμαστε ξεκάθαροι. Ιδίω ό,τι φορά την παράγραφο 5, η εξολογήση αντικτύπου εξάντια της Επιτροπής καλύπτει οικονομικές ε, κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ πτυχέ των συμφωνιών και από το 2011 και μετά καλύπτουν και στοιχεία που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρξε μια συζήτηση για τι αξιολογήσει αντικτύπου. Η γνώμη τη Επιτροπή είναι ότι το αποτέλεσμα αυτών των αξιολογήσεων είναι ε, εύρωστο και τεκμηριωμένο. Οι βιώσιμε αξιολογήσει αντικτύπου διεξάγονται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και συνεχίζονται και μετά. Είναι χρήσιμε και διευκολύνουν κάτι που έθιξαν πολλά μέλη. Η μεγαλύτερη προβολή μας και εξωστρέφεια. Κλείνοντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αφοσιωμένη στην ε, διατήρηση ε, των σχέσεών της με την ε, κοινωνία των πολιτών. Καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες για να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών. και αν θέλετε και για του ορισμού τη εμπορικής Πολιτική μπορούμε να τα εξετάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο εισηγητή, συμπερασματικά. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο γιατί συνειδητοποιώ ότι ξεκινήσα μία νέα διαδρομή σε ένα εξερευνητό έδαφος ίσως. Φυσικά και θα λάβω υπόψη όλα τα σχόλια. Τώρα, μια μερική απάντηση η εξολογηση ξεκινήσει από δύο σημεία. Καταρχήν, το θέμα της δημόσιας διαβούλευσης. Πολλές φορές συνειδητοποίησα ότι η Κομισιόν θεωρεί ως ισχύουσα μια δημόσια διαβούλευση όπου έχουν συμμετέχει μόνο δύο-τρία κράτη-μέλη και με ένα πολύ περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Από τη δική μου σκοπιά αυτό αποτελεί μια δύσκολη βάση να στηριχτεί κανείς. Επομένως η πρότασή μου να διευρυνθεί η βάση της αφετηρίας ε, ίσως θεωρώντας ως ισχύσεις μόνο τις δημοσίες διαβουλεύσεις όπου έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή θα μπορούσε να είναι μια λύση για το άλλο θέμα της αγγλικότητας και της ρήτρας διασφάλισης. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα ότι οι αρμοδιότητες της εμπορικής πολιτικής πρέπει να είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα διαφορετικό βάρος ε, στις εμπορικές πολιτικές των κρατών μελών. Όμως συνειδητοποιώ ότι και στα 28 κράτη-μέλη υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις γιατί διαφέρουν πολλοί χώρες μεταξύ τους και επομένω η δυνατότητα κάποιο κράτος μέλος να μπορεί να ενεργοποιήσει ρήτρε διασφάλισης, δηλαδή εν μέρη να τροποποιήσει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαφυλάξει μια δική του ιδιαιτερότητα της αγοράς, νομίζω ότι είναι κάτι ευκταίο. Φυσικό θα τα λάβω υπόψη όλα αυτά και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και στο μέλλον για το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ. Η, η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 20 Μαΐου 12 το μεσημέρι. High noon. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 9. Θυμάστε ότι ε, αντιστρέψαμε τα δύο θέματα το περίφημο θέμα, θέμα της κλωνοποίησης. Ε, καμιά φορά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κλωνοποίηση και για τα μέλη εδώ, αλλά δεν υπάρχει ακόμη. Και η, η δική μας είναι η κυρία Ντάλινγκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτά, γιατί αλλιώς θα μπορεί να γίνουμε και περιττοί. Είναι η δεύτερη φορά που το εξετάζουμε στην, στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τη συνεισφορά τους και για τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Και στην τελευταία συζήτηση στην Επιτροπή ε, είχα παρουσιάσει επιθέσεις των σοσιαλιστών. Θα επικεντρωθώ λοιπόν στις 15 τροπολογίες που έχουν από κατατεθεί από άλλα μέλη που καλύπτουν ουσιαστικά τέσσερις ε, θεματικές ομάδες. Θα ήθελα να διατρέξω λοιπόν τομή αυτά τα ζητήματα. Αρχικά, σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα της απαγόρευσης, κάποια μέλη πρότειναν να γίνει μόνιμη και όχι προσωρινή απαγόρευση. Κατανοώ ότι αυτή η προσέγγιση στερίζεται και από ε, την καθέληνα αρμόδια επιτροπή. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τις σκέψεις ε, των συναδέλφων. Για τους σοσιαλιστέ, το κύριο σημείο είναι να υπάρχει ρήτρα αναθεώρηση στην νομοθεσία ανεξαρτήτως της φύσης τη της ούτω ώστε να μπορεί να υπάρξει μελλοντική επαναξιολόγηση. Δεύτερον, η νομική μορφή της πρότασης. Η πλειονότητα στηρίζει το κείμενο να γίνει κανονισμό και όχι οδηγία. Οι συνάδελφοι στην ΕΝΒΗ και σε άλλες επιτροπές ε, ασχολούνται και πάλι με αυτή τη βάση. Δεν ε, μας δημιουργεί πρόβλημα η ενσωμάτωση αυτών των ε, τροπολογιών, αλλά να ακούσουμε και τις απόψεις. Μετά, δύο εφαρμογή. Ορισμένα μέλη πρότειναν να διευρυνθεί ο κατάλογος των ζώων, ενώ άλλοι θέλουν να περιοριστεί ο κατάλογος των ορισμών στα αστροδίου, ό,τι αφορά τον απολογικό υλικό και τους απογόνους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι οι άλλες επιτροπές θέλουν να ακούσουν και τη δική μας γνώμη σε ό,τι αφορά το, ε, τους κανόνες που συνδέονται με το διεθνές εμπόριο. Εμείς πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ληφθούν αναλογικά μέτρα βάσει της ευημερίας των ζώων ε, και στοιχείων ηθικού προβληματισμού και να είναι όλα αυτά συμβατά με τον ΠΟΕ. Και θα πρέπει να αποδυναμώσουμε αυτό το μήνυμα με το να έχουμε δυσανάλογα μέτρα. Από αυτήν την άποψη θα ήθελα να ακούσω τις ε, απόψεις των ε, συναδέλφων και η τροπολογία 48 μπορεί να αποτελέσει ε, τη βάση ενός καλού συμβαστικού κειμένου. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ειχνηλασιμότητα, υπάρχουν παρατηρήσεις που έγιναν από πολλούς, ALDE, EFDD και GUE, είναι σημαντικά τόσο ανέφεραν. Ζητούμε διατάξει συναλυσιμότητα από του εμπορικού εταίρου. Μπορεί να μην είναι δυνατό κάτι τέτοιο ε, σε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό. Όμω, ίσω θα μπορούσαμε να βρούμε μία διατύπωση για να συνδέσουμε αυτά τα στοιχεία με τι συνεχιζόμενε διαπραγματεύσει ε, και ε, το πλαίσιο SPS του ΠΟΕ. Θα μπορούσαμε αυτά να τα ενσωματώσουμε στο κείμενο της νομοδότησης. Αυτά είναι τα τέσσερα κύρια σημεία ε, για τα οποία κατατέθησαν ε, τροπολογίες. Έχουμε και συνάντηση των σχεδόν την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να ακούσω τις γνώμες σας σήμερα και θέλω να ε, συνεργαστούμε επικοδομητικά όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχουν οι σκιώδεις. Ο κύριος Φίζας πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την συγγήτρια για το έργο της. Πάντοτε έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία σε όλες τις περιπτώσεις. λοιπά, στην Ιγυρία σε μια εκλογική αποστολή κατά την ε, ανταλλαγή απόψεων ε, ο κ. Κασπάρη είχε πει και είναι γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι είναι κατάλληλη η τοποθέτηση της εισηγήτριας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες για να δεχτούμε την πρότασή της και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εργαστούμε ε, τόσο καρποφόρο όπως κάναμε και για το Nobel Food. Μία δροπολογία έχω να προτείνω και προτείνω να αλλάξουμε από την οδηγία και να έχουμε κανονισμό. Αυτό συνάδει και με όσα θέλουν οι συγγητές από τις Επιτροπές Άγκρη και Ένβη. Και επίση νομίζω ότι είναι σκόπιμο να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω κανονισμού για να αποφύγουμε διαφορές στην εφαρμογή που θα μπορούσαν να στρεβλώσουν το εσωτερικό εμπόριο και να έχουν άνοιξο αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο με τρίτους ο συνάδελφος Αλντο Πετρετσελό έχει παρουσιάσει μια τροπολογία που δεν μας θέτει κανένα πρόβλημα. Τώρα, για τις τροπολογίες που έχουν κατευθεί από άλλες ομάδες πρέπει να τις μελετήσουμε λεπτομερώς, αλλά θέλω να αναφέρω το εξής. Συμφωνώ στο να απαιτηθούν τα ίδια μέτρα που ζητάμε και από τους κτηνοτρόφους, δηλαδή να απαιτήσουμε τα ίδια και από τις τρίτες χώρες από όπου εισάγουμε κρέας Φυσικά όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Επίση, νομίζω ότι είναι λογικό να συντάξουμε μια νομοθεσία που να μπορέσουμε να τη θέσουμε σε εφαρμογή, να είναι ρεαλιστική. Και Ξεκινώντα από αυτέ τι δύο προποθέσει, θα ήθελα η Κομισιόν που είναι παρούσα εδώ να μα πει την άποψή τη για την δυνατότητα ε, δημιουργία ενό συστήματο ανιχνευσιμότητα για τα κλωνοποιημένα ζώα, του απογόνου του και για το αναπαραγωγικό υλικό. Γιατί, επαναλαμβάνω, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο νόημα να θεσπίζουμε μέτρα, αν στη συνέχεια δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Επομένως, θα ήθελα να δω και ποια είναι η άποψη της Κομισιόν σχετικά με το ζήτημα αυτό. Και φυσικά στην Εδρία των σκιωδών θα έχουμε και την δυνατότητα να εμβαθύνουμε περαιτέρω σε όλα αυτά τα σημεία. ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ. Ήδη ευχαρίστησα την συγκεκριτή στην πρώτη εντέλεγη απόψεων ε, πριν ένα μήνα περίπου και αφού συμμετείχα ως μέλος της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος στην κοινή συνεδρίαση που είχαμε στη βασική συνάντηση και άκουσα μία σειρά επιχειρημάτων ε, και κάποια ήταν ε, και ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένα για το θέμα αυτό και ε, μπορώ να πω ότι υπήρχε και μια σπαστική προσέγγιση από την κυρία μου και την κυρία Μόη που μένω ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια για την πολύ ισορροπημένη χρηματοδότηση που μας παρουσιάζει εδώ το είχα ήδη πει, αλλά το αναφέρω και πάλι εδώ και φαίνεται και από τις τροπολογίες μου. Επερασπίζει τρεις αρχές ε, που είναι σημαντικές για τους φιλελεύθερους και ζήτησα το προσωρινό χαρακτήρα, ε, μάλλον συγγνώμη, η τροπολογία για τον προσωρινό χαρακτήρα, δεν υπάρχει πλέον, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ε, φυσικά η τεχνική δεν λειτουργεί και είπαμε ότι δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σήμερα στο θέμα αυτό. Έχουμε πραγματικά ψυχικά προβλήματα, τα ζώα υποφέρουν, όμως εμείς αρνούμαστε να ε, ταχθούμε κατά της πρόοδου ως φιλελεύθεροι και φυσικά θέλουμε και την παρέκκληση στην εξαίρεση από την κλωνοποίηση που θα γίνεται για ε, λόγους έρευνας, για να προστατευτούν τα σπάνια είδη ή για την έρευνα για τα φάρμακα. Η τροπολογία 22 ελπίζω να υποστηριχτεί. Η τρίτη αρχή πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας υπόθηκε επίση ε, είναι να σεβόμαστε τις απαγορεύσεις ε, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Επίσης, Θέλω να ε, κάνω και μια σημαντική διαφοροποίηση, δηλαδή είναι η θέση σας να έχουμε απαγόρευση για όλες τις γενιές των απογόνων. Εγώ προτείνω στις τροπολογιες K42-46 αυτή η απαγόρευση να ε, καλύπτει την πρώτη γενιά, τους άμεσους απογόνους ε, και θέλω να δηλώσω και ότι λυπάμαι για το ότι η Κομισιόν ε, στην αρχή της πρόταση να αποφύγει τη συζήτηση για τους απογόνους ε, και έχουμε δει με όλες τις συζητήσεις που κάναμε ότι γύρω από το θέμα των απογόνων επικεντρώνονται οι συζητήσεις μας. Ένα άλλο θέμα, λιγότερο επίμαχο, το αναφέρω και ο προηγούμενο ομιλητή. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπερασπίσω τι τροπολογίε του, είτε να περάσουμε από οδηγία σε κανονισμό, είτε να καλύψουμε και άλλα είδη ζώων, ε, αν εφαρμόζεται η τεχνική της κλωνοποίησης, αλλά ήδη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να κλείσω προς την Κομισιόν, αν ε, λάβουμε υπόψη το status quo, του status quo, που μας είχε αναφέρει και στην πρώτη ανακοίνωση ε, το 2010. Θα έλεγα ότι αυτό το status quo δεν βοηθά σε μια προσέγγιση στην οποία ελπίζουμε να φτάσουμε μια μέρα σε μια προσέγγιση των θεσεών μας. Στην προηγούμενη συζήτηση η Κομισιόν είχε πει ότι μία μελέτη για την ε, ετικετοθεσία των κλωνοποιημένων ζώων και των απαγωνών τους γίνεται αυτή τη στιγμή από τη ΓΔΑ η μελέτη αυτή θα δημοσιευτεί πριν από την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει τον Ιούλιο. Και δεύτερη ερώτηση, θεωρείτε ότι αυτή η ετικετοθεσία ε, είναι κάτι που μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή και αν ναι, γιατί η Κομισιόν, και το άκουσα αυτό σε προσφατή ακρόση, συνεχίζει να θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η εχνηλασιμότητα Έχω ένα έγγραφο της Κομισιόν εδώ το 2010 που αναφέρει ότι θεωρείται ότι είναι appropriate αυτό. Κατάλληλο έτσι λοιπόν πώς το 2010 θεωρούσε την χρησιμότητα κάτι σκόπιμο ενώ σήμερα θεωρεί η Κομισιόν ότι είναι δυσανάλογη και ότι δεν ε, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Εδώ στην Επιτροπή ΙΝΤΑ όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε έναν εμπορικό πόλεμο με τις τρίτες χώρες, αλλά επίσης για μας και υπενθυμίζω ότι αυτή είναι η θέση των φιλελευθερών παρά ε, το ότι εδώ φαίνεται εμείς να παρακλίνουμε κάπως σε μια κατά τα άλλα ομόφωνη θέση που παρουσιάζεται από τους εμείς δεν θα, θέλουμε, δεν θα θέλαμε να γίνει και το οτιδήποτε που θα σημαίνει ότι θα έχουμε μείωση των προτύπων μας. Τώρα για τους συντηρητικού και ελεύθερους, ο κύριος Ζαχράντιλ. Ευχαριστώ, εκπροσωπώ τον κύριο Μπιέχ και είναι μας. Η ομάδα μας έχει υποβάλει μία τροπολογία, όπου καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει την πρόταση. Ανησυχούμε για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο. Τα εξή. Πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και να δημιουργήσει προβλήματα, ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ και τις χώρες του Mercosur, όπου υπάρχει ελεύθερο εμπόριο κλωνοποιημένων ζώων. Υπάρχουν και άλλοι εμπορικοί μας εταίροι που έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες σε σχέση με τη συμβατότητα όλων αυτών με τον ΠΟΕ, Καναδάς, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αργεντινή, Αυστραλία, Αργεντινή. Άρα μπορούμε να έχουμε προβλήματα εδώ, ζημίες. Και τρίτον, υπάρχει το θέμα της ίχνη λασιμότητας και των ε, εξετάσεων. Η χνηλασμότητα μπορεί να δημιουργήσει υψηλό κόστος για τους ε, παραγωγούς τροφίμων και τους γεωργούς και για τις εξετάσεις και τα τεστ δεν ξέρουμε αν υπάρχει τεστ αυτή τη στιγμή που να μπορεί να ξεχωρίσει μεταξύ κλωνοποιημένων και μη ζώων και ζωικών προϊόντων. Θεωρούμε ότι υπάρχει επαρκή νομοθεσία ήδη. Η νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα που θα διασφάλιζε ότι δεν είναι δυνατόν ε, να υπάρξουν τέτοια τρόφιμα στην αγορά χωρίς τους απαραίτητους πρώτερους ελέγχους. Άρα θεωρούμε ότι αυτή η νομοθεσία στέλνει μάλλον αντικό μήνυμα για την έρευνα, την απασχόληση και την επιστήμη και θα μπορούσε να αποθαρρύνει και επενδυτές να επενδύσουν στην Ευρώπη. Προτείνουμε λοιπόν να απορριφθεί αυτό το σχέδιο πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Μινά. Ευχαριστώ. Διαβάζω το κείμενο από την ε, σκιώδη μας Ελεονόρα Φορέντσα Ευχαριστώ πρώτον ε, την εισηγήτρια για την εργασία της που πηγαίνει προς την διακατεύθυνση που και εμείς θεωρούμε πως είναι αναγκαία για το θέμα αυτό. Τονίζουμε τα βασικά στοιχεία που για μας θα πρέπει να προσθεθούν για να ενισχύσουν την απαγόρευση ε, εμπορίου κλωνοποιημένων ζωικών προϊόντων. Η σήμανση είναι πολύ σημαντική γιατί πολλές τρίτες χώρες ήδη τη χρησιμοποιούν για να επίσης είναι αναγκαία υποχρεωτική ηχθυλασιμότητα. Διότι αλλιώς αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Αν δεν μπορούμε να έχουμε και για το σπέρμα και για τα προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τώρα συζητάμε το TTIP με τις ΗΠΑ που επιτρέπει την κλωνοποίηση για την παραγωγή τροφίμων. Ένα από τα ζωτικά σημεία, τα κρίσιμα σημεία της ε, διαπραγμάτευσης είναι πώς θα διασφαλίσουμε το σεβασμό της αρχής της πρόληψης, βασική αρχή για την πολιτική τροφίμων μας. Εκτιμούμε την εργασία της εισηγήτριας, αλλά πραγματικά ελπίζουμε η γνωμοδότηση αυτή να βέλτιωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, και ο Πρόεδρος και η κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ εδώ θέλω να θέσω μια ερώτηση στους συναδέλφους, να ρωτήσω αν εσείς θα δίνετε στα παιδιά σας γάλα από κλωνοποιούν ζώο ή το κρέας τους. Γιατί αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε ότι είναι σίγουρα αυτά τα προϊόντα, γιατί δεν υπάρχουν μελέτες και δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει με την κατανάλωση τέτοιων κλωνοποιημένων προϊόντων, προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα. Σε 20 χρόνια μάλλον θα έχουμε αυτές τις μελέτες, αλλά μέχρι τότε θα είμαστε δημιουργημένοι εμείς. Το κλωνοποιημένο ζώο είναι ακριβώς γενετικό αντίγραφο και αν ένας κτηνοτρόφος δει ότι δίνει περισσότερο κρέας, φυσικά θα θέλει και τα υπόλοιπα ζώα να δίνουν την ίδια παραγωγικότητα. Γιατί φυσικά θα θέλει ε, ακριβώς να έχει και προβληψιμότητα. Σε αυτό το σημείο αναρωτιέμαι ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ζώου και ενός αυτοκινήτου και αν ε, ίσως αυτό θα μπορούσε να εκτιμηθεί από μια σκοπιά εντελώς ε, οικονομική. Νομίζω ότι ε, υπάρχουν ερωτηματικά που πρέπει να θέσουμε ήδη. Χρησιμοποιούμε τη φύση όπως θέλουμε και χρησιμοποιούμε τα ζώα για να εξυπηρετήσουμε την διατροφική βιομηχανία. Εδώ όμως ξεπερνάμε κάθε φαντασία. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα δεινά στα ζώα, μόνο ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό ε, των κλωνοποιημένων ε, εμβρίων γεννάται ζωντανό ε, και βέβαια κινδυνεύουμε να χαθεί και η βιοπικιλότητα και η γενετική διαφοροποίηση έκθεση. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν λέει τίποτα για τους απογόνους των κλωνοποιημένων ζώων. Έτσι λοιπόν μπορούμε να επιτρέψουμε τις πρακτικές, μπορούμε να επιτρέψουμε να υποφέρουν τόσο τα ζώα. Εγώ θα έλεγα όχι. Και όσο αφορά το έργο της Επιτροπής, ε, λέγω ότι θα πρέπει να ε, προσέχουμε όχι μόνο το εμπόριο των κλωνοποιημένων ζώων, αλλά και των ζωντανών ζώων και του γενετικού του υλικού. Έχουμε πάρα πολλού λόγου και ηθικούς. Ε, δεν γνωρίζουμε δυστυχώς τις συνέπειες μιας μακράς κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων. Εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε και σύστημα ειχνηλασιμότητας και αντικαιτοσίας και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με την TTIP γιατί ελπίζω τουλάχιστον εκεί που δεν θα αρκεί η δουλειά του νομοθέτη να αρκέσει η κρίση του καταναλωτή. Εδώ ε, Δυστυχώ πρέπει να πω ότι η πρόταση τη Κομισιόν είναι πολύ αδύνατη και πιστεύω ότι αυτό θα διευκολύνσει τη σχέση σε ισχύ της TTIP. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να μα λέει ότι δεν θα επηρεάσει ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά ήδη αλλάζουμε του νόμου αυτού επομένω κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Φλου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Σημείωσα κάποια σημεία, είχαμε κάποια σχόλια που στράφηκαν προς την Κομισιόν, η χρησιμότητα είναι σκοπός. Να πω καταρχήν δύο λόγια για το πεδίο εφαρμογή ε, όταν ε, έκανε την πρόταση της η Κομισιόν. Δεν είχαμε λάβει υπόψη όλα τα είδη. ότι η τεχνολογία δεν τα καλύπτει. Έτσι λοιπόν έχουμε αναφερθεί μόνο στα είδη που τα θεωρήσαμε σχετικά. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή ε, και στους απογόνους. Τώρα μιλάμε μόνο για τα κλιμαπημένα ζώα αυτά καθ' αυτά. Το να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή και στους απογόνους θα σήμαινε ότι δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε τα μέτρα που αφορούν την ευημερία των ζώων και έχει προσδιοριστεί από την ΕΦΣΑ, όπου βασίσαμε και την πρότασή μας. Γιατί θεωρούμε ότι οι απόγονοι των κολομπημένων ζώων ε, ε γίνονται περνούτος χάρη με τεχνητή γονιμοποίηση και θα πρέπει να αιτιολογούνται με άλλους λόγους, λόγω ηθικών ανησυχιών, το χάρη. Έχουμε επιφυλάξεις λοιπόν σε σχέση με τη διαβρύση του πεδίου εφαρμογή, ιδίω για τους απογόνους των κλωνοποιημένων ζώων. Και επίσης ε, αναφέρθηκε και θέμα ασφάλειας από την τελευταία μιλήτρη η ΕΦΣΑ με σαφήνεια μας έχει πει ότι η κλωνοποίηση δεν είναι θέμα διατροφικής ασφάλειας, δεν υπάρχει κίνδυνος. Επίσης, θα επανέλθω σε ένα θέμα που τέθηκε πολλές φορές, στην ειχνηλασιμότητα. Και εδώ σημείωσα διάφορες απόψεις. Η κυρία Ρης ανέφερε τη θέση της Κομισιόν του 2010 και τη σημερινή θέση της Κομισιόν. Από το 2010 έχουμε επιτελέσει μια μελέτη αντικτύπου που αποτέλεσε τη βάση για τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει. Και αυτή η μελέτη αντικτύπου σχετικά με την ε, δυνατότητα και θεσίας και επιβολής ε, κανόνων για τα κλωμμένα ζώα και τους απογόνους απέτυχε στο τεστ αναλογικότητας γιατί θεωρήθηκε ιδιαίτερα πολύπλοκη και δαπανηρή. Η κυρία Ρεής αναφέρθηκε σε μία μελέτη η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν, σωστά. Τώρα, εξετάζουμε αυτό το θέμα της αποτυχίας του τεστ αναλογικότητας λόγω των δαπανών και του κόστους. Κομισιόν κίνησε μια μελέτη για να το απελευθεύσει αυτό και η μελέτη αυτή θα είναι διαθέσιμη, έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2015. με Αυτό νομίζω απάντησα στα κυρία θέματα που τέθηκαν. Υπήρχαν κάποια νομικά ζητήματα, αλλά δεν θα ήθελα να μπω στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Η Τζουντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους σκιώδες. Νομίζω ότι έχουμε τη βάση για έναν ευρύ συμβιβασμό και θα μπορούσαμε να βρούμε λύσεις στις συναντήσεις των σχεδόν συγητών την επόμενη εβδομάδα. Και εκτιμώ είπαν οι συνάδελφοι ποια είναι τα κύρια σημεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε όσο την αποτελεσματικά τη συνάντηση των σκιωδών με την εξαίρεση μιας ομάδας από ό,τι φαίνεται μπορούμε να βρούμε ένα είδος συμβιβασμού ως προς το να τροποποιήσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας και τα σχόλια και υπομονώ για τη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ, να σας υπενθυμίσω ότι φυσικά θα πρέπει να μείνουμε εντός των αρμοδιοτήτων μας. Έτσι, λοιπόν να ε, ξέρω αν θα μπορούσαν ε, όλοι οι συνδεσμοί να περάσουν, να το έχετε κατά νου. Ψηφοφορία 28 Μαΐου. Σας ευχαριστώ. Και φτάνουμε τώρα στο αρχικό σημείο 8 για τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα μη γεωργικά προϊόντα. Ξέρετε, υπό το καθεστώς του τρίψ είναι δυνατόν αλλά έχουμε ένα κανονισμό μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα γεωργικά προϊόντα. Και τώρα η συζήτηση είναι ότι ορισμένα από τα κράτη-μέλη έχουν ορισμένες νομοθεσίες ε, για τα μη γεωργικά προϊόντα και αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κυρία Μόσκα. Ναι, σας ε, ευχαριστώ που αλλάξατε και το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ήταν απαραίτητο γιατί ήμουν απασχολημένη σε άλλη επιτροπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ε, δουλειά που κάναμε με τους σκιώδεις εισηγητές για την γνωμοδότηση αυτή. Πραγματικά ήταν πολύ επικοδημοτικό το κλίμα. Και αυτό μου οδηγεί να πω ότι την επόμενη συνάντηση, στην επόμενη συνεδρία στον Ιούνιο, θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την γνωμοδότηση. Όπως είπαμε και στην περασμένη συνεδρίαση, αυτή είναι μια γνωμοδότηση που η δική μας ε, Επιτροπή κλήθηκε να χορηγήσει στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια καθήλυντα Επιτροπή. Εγώ προσπάθησα να αναφέρω και να συλλέξω εδώ κάποιες ενδείξεις ε, που αναφέρθηκαν στην ε, συζήτηση της περασμένης φοράς. Εκεί Είχαμε ήδη δει διαθεσιμότητα να υποστηριχθεί η υπόθεση να διευρυνθούν οι γεωγραφικές ενδείξεις και σε μη γεωργικά προϊόντα. Περιορίζομαι λοιπόν στο να αναφέρω τα κύρια σημεία της γνωμοδότησης που πιστεύω ότι μπορεί να είναι αυτά επί των οποίων η Επιτροπή μας ε, έχει νόημα να εκφραστεί θεωρήσαμε σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι με μια ad hoc ε, νομοθέτηση θα ήταν πολύ πιο σκόπιμη γιατί και θα προστατεύαμε τον καταναλωτή αμυντικά αλλά θα είχαμε και επιθετικά συμφέροντα για να βελτιώσουμε την παρουσία των προϊόντων και να εγγυηθούμε τον θεμητό ανταγωνισμό. Δεύτερον, τα κράτη θα πρέπει να βρουν μια πολιτική συμφωνία ε, που ουσιαστικά να μπορεί να δίνει τεχνικές δυνατότητες για να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να διευρύνουμε το μηχανισμό προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και σε άλλα προϊόντα. Και έχουμε υπογραμμίσει μία από τις αντισυχίες που ανέκυψαν από την συζήτηση της προηγούμενης φοράς, δηλαδή την αναγκαιότητα οι μηχανισμοί αυτοί να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικοί αλλά και όσο δυνατόν λιγότερο δαπανηροί και από οικονομική σκοπιά και από γραφειοκρατική σκοπιά, έχοντας κατά νου ότι κύριοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι και η παραγωγή αλλά και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Στη συνέχεια εντοπίσαμε την αναγκαιότητα να υπογραμμίσουμε πως τα σημερινά πρότυπα προστασία θα πρέπει να θεωρηθούν ως σημείο αυθεντηρίας για μελλοντική επέκταση. Γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αμφισβητήσουμε τα σημερινά επίπεδα προστασία εξ ονόματο μια μελλοντική δράση, που δεν είναι και βέβαιη. Το σύστημα προστασία γεωγραφικών ενδείξεων, γεωργικών προϊόντων λειτουργεί αποτελεσματικά και πιστεύουμε ότι μπορεί να θεωρηθεί ω μοντέλο για μια πιθανή επέκταση του μηχανισμού σε μη γεωργικά προϊόντα. Ένα σύστημα ε, θα συνεκτικό θα μπορούσε να διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, διαπραγματεύεται διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και αναγνώριση και στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Επομένως, η εσωτερική συνοχή θα ήταν χρήσιμη σε ό,τι αφορά το πώς προδεύουν οι συζητήσεις ε, και σε πολυμερές επίπεδο είναι δύσκολο να είμαστε αξιόπιστοι ε, συνομιλητές αν δεν υπάρχει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνία. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Κομισιό να οθήσει τα μεμονωμένα κράτη-μέλη να επικυρώσουν το πρωτόκολλο της Λισαβόνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Θεωρούμε ότι επίση είναι σκόπιμο η Κομισιόν να δεσμευτεί για να εισαγάγει ένα κεφάλαιο για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία στι διαπραγματεύσει που υλοποιούνται σήμερα αλλά και στο μέλλον και να δοθεί ιδέουσα προσοχή στο θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων και σε ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο ελπίζουμε ένα σύστημα προστασία του που θα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για, κατά την άποψή μα, θα ήταν προτιμότερο από την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων, γιατί αυτό θα διευκόλυνε το να ξεπεράσουμε τις διάφορες αποκλήσεις που υπάρχουν σήμερα. Και τέλος, είναι σκόπιμο υπό ε, την οπτική της ανακοίνωσης για την στρατηγική της Κομισιόν για την εμπορική πολιτική να αναφέρεται με σαφήνεια ένα σημαντικό ρόλο στην πρόθεση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτή είναι μια σύνθεση της γνωμοδότησής μας και ελπίζω να συμφωνήσετε ευρέως. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ως και του έλκο, ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρία Συγγήτρια, αγαπητά φίλοι. Η συνάδελφος Τάκα Σαϊφή, τελευταία στιγμή μου είχε ένα κόλλημα, μου ζήτησε να μεταφέρω τα λόγια της. Θα σας αναγνώσω λοιπόν τη δήλωση που ήθελε να κάνει. Ήθελα αρχικά να συγχαρεί την κυρία Τροσφαγιά το σχέδιο γνωμοδότησή τη, ιδίω ό,τι αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν γέννη, Συμμεριζόμαστε τις ε, θέσεις που εκφράζει η κυρία Μοσκάρ στην, ε, στο κείμενό τη. Είναι σημαντικό όμω να αναγνωρίσουμε ότι αυτέ οι προεκτάσει θα πρέπει να επιτρέψουν την προστασία των επιχειρήσεων και των πολιτών μα από το παρεμπόριο και τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και θα επιτρέψει αυτό να ενισχύσουμε την θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι εμπορικέ και διεθνεί ε, διαπραγματεύσει. Τα είπαμε αυτά και σήμερα το πρωί για την επίσκεψή μα στο Βιετνάμ. Όπω έχουμε ήδη αναφέρει στην πρώτη ανταλλαγή απόψε, η παράγραφος 4 μιλά για αναγκαιότητα θέσπιση ε, απλών διατάξεων ε, με χαμηλό κόστος και χαμηλό επίπεδο δέσμευση σε ό,τι αφορά τα μη γεωργικά προϊόντα και στι γεωγραφικές ενδείξεις. Συμφωνούμε με αυτό το αίτημα και υπογραμμίζουμε την ανάγκη ενό χαρακτηριστικού για ένα σύστημα το οποίο θα είναι κυρίω ε, προσβάσιμο από μικρομεσαίε επιχειρήσει. Τέλο, ό,τι αφορά τι πολυμερεί ε, ε, στον ΠΟΕ, Χρειαζόμαστε περισσότερη στήριξη για τα μη γεωργικά προϊόντα, ιδίω σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει ε, για τα αντεπεσέ. Κινούμαστε στην κατεύθυνση του αρχικού κειμένου. Θέλουμε να συμπληρώσουμε τις επιμέρους παραγράφους ε, του σχέδιου γνωμοδότηση και θα ήθελα προσωπικά να επισημάνω ότι για μένα αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί αρχικά διευρύνουμε ε, τα ζητήματα αυτά στα μη γεωργικά προϊόντα και μετά εξετάζουμε και την οικονομική και την πολιτιστική κληρονομιά ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Et maintenant... Ευχαριστώ. Η κυρία Σαντσάουερ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότησης. Εκτιμώ την ποιότητα του έργου της ε, που επισημαίνει και τα ωφέλη ε, για την εσωτερική αγορά και για τις εμπορικές μας σχέσει στο εξωτερικό. Αναμφίβολα, ο σκοπός της ε, οι στόχοι μάλλον υπονομεύονται τη εσωτερική αγορά με τι γεωργικέ ενδείξει για τα μη γεωργικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη δει την επιτυχία τη διασφάλιση ποιότητα και Προέλευση από ένα σύστημα για τα γεωργικά προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να επεκταθεί αυτή η προστασία, ενώ η παραδοσιακή εθνική προστασία επαρκεί για κάποιες μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνοριακές συναλλαγές, Παρ' αυτά αυτό το σύστημα είναι πολύ σημαντικό μειονέκτημα για τους εξαγωγείς και γενικά τις επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα σε παραπάνω κράτη-μέλη. Υπάρχουν και κάποια κύρια σημεία που θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, ένα παράλληλο σύστημα προστασίας. Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας δεν σημαίνει την απαλυφή της προστασίας σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν ενδιαφέρονται όλοι οι παραγωγοί να λάβουν προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως αν δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα κράτος μέλος. Το ενιαίο αυτό σύστημα θα πρέπει λοιπόν να συνεπάρξει με τα εθνικά συστήματα, ώστε οι παραγωγοί να επιλέγουν τον τύπο προστασία που ε, θεωρούν ότι του ε, ταιριάζει καλύτερα. Δεύτερον, είναι επίση σημαντικό να προσδιορίσουμε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί μία ε, προσέγγιση ανακλάδο, κάτι που έχει ήδη εφαρμοστεί για, τα, για τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα γεωργικά προϊόντα. Ήταν δύσκολη κατάρτιση καταλόγων και μη αποτελεσματική. Για λόγους αποτελεσματικότητας λοιπόν αυτό το μελλοντικό ε, σύστημα θα πρέπει να, να είναι οριζόντιο και να καλύπτει όλες τις, τις κατηγορίες. Τέλος, ε, δεν θα πρέπει να υπονοούμε και να υποτιμούμε την ανταλλαγή πληροφοριών. Η προστασία ευρωπαϊκού συστήματος μπορεί να έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο, όμω για να αποφεληθούν όλοι από αυτές τις διατάξεις, οι πληροφορίε θα πρέπει να φτάνουν μέχρι τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Ευχαριστώ πολύ και προβλέπω και σε μελλοντική συνεργασία ε, για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ να διαβάσω ένα κείμενο της Λεωνόρα Φορέντσα. Ευχαριστούμε τον Σίτη η επέκταση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων, εάν θα ενθαρρύνει την πληροφόρηση για τους καταναλωτές και την διαφάνεια και θα προβάλλει και τους παραγωγούς, είναι κάτι θετικό. Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι ένα μέσο για υψηλότερη προστιθέμενη αξία προς συγκεκριμένε περιοχές και να δημιουργήσει στενότερη σχέση με τους καταναλωτές μέσω σαφών κανόνων για προϊόντα ποιότητας. Προτεραιότητες θα πρέπει να είναι ένα σύστημα ενωσιακό προστασίας που δεν θα αποτελέσει μείωση των προστασιών που ήδη δίδονται σε εθνικό επίπεδο αλλά που θα αξιοποιήσει τις ε, καλύτερες διατάξεις για την ίχνη λασιμότητα, την υπεράσπιση των επιπέδων ε, παραγωγής και απασχόλησης. Πρέπει να ενισχυθεί αυτή η γνωμοδότηση στα εξή δύο σημεία για την επίπτωση στο παγκόσμιο εμπόριο. Πρώτον, η επίπτωση της επέκτασης σε συμφωνίες ελευθερού εμπορίου, ιδιαίτερα στο TTIP, όπου η ζήτηση ε, θεμάτων γεωγραφικών ενδείξεων δημιουργεί πολλές διαφωνίες. πάντα θεωρούσαμε ότι το TTIP μπορεί να, αδυναμώ, να αποδυναμώσει το σύστημα γεωγραφικής, γεωγραφικών ενδείξεων που έχουμε. Οι ΗΠΑ το θεωρούν εμπόδιο στο εμπόριο. Ενώ εμείς θεωρούμε ότι είναι προστασία των τοπικών παραδόσεων είναι των μεγάλων πολυεθνικών. Βλέπουμε να υπάρχει ενδεχόμενο διαφωνίας μεταξύ της δικής μας βούλησης να ενισχύσουμε αυτό το σύστημα και τη διαπραγμάτευση ε, μια συμφωνία που μπορεί να αποδυναμώσει. Αυτή είναι μια αντίφαση και θα την τονίσουμε. Δεύτερη προτεραιότητα. Δίκαιη πρόσβαση για το σύστημα αυτό από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα τις πιο φτωχές, ιδιαίτερα μέσα αναθεώρησης του άρθρου 23 του TRIPS. Θεωρούμε ότι η προτεραιότητα του συστήματος, της επέκτασης του συστήματος αυτού πρέπει να είναι να προστατεύσει όλους τους παραγωγούς παντού στον κόσμο, ιδιαίτερα μικρούς παραγωγούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Έξι έχουν στήσει τον λόγο και μας έχουν μείνει μόνο δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ να είστε ως δυνατόν ε, ταχύτεροι. Ο κύριος Ζαχράντιλ. Θα διαβάσω κι εγώ τώρα ένα κείμενο της Εύα Μακλάρκιν Ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρεθεί. Δεν είναι ακόμη πεπισμένο ότι χρειάζεται να επεκταθεί σε μη γεωργικά προϊόντα. Θα προτιμούσε η Επιτροπή να κάνει μια πλήρη μελέτη αντικτύπου για το τι ωφέλη θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις μας. Μια τέτοια μελέτη θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε και τι τύπου επέκταση θέλουμε για μη γεωργικά προϊόντα. Γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα μεν από τα δε. Η επέκταση του ιδίου συστήματος είναι υπεραπλούστευση. Και πρέπει να συμβάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να καταλάβουμε κατανοεί τη σημασία της προστασίας της ποιότητας των προϊόντων που επιζητούνται παντού από τις χώρες μας, θα θεωρούσα ότι οι νόμοι για τα σήματα κατά τεθέν επαρκούν. Το σύστημα αυτό είναι σε εξέλιξη, γιατί αυτό το σύστημα σημαίνει ότι και οι καταναλωτές ε, γνωρίζουν τα προϊόντα ποιότητας και υπάρχει αυστηρή προστασία των γεωγραφικών περιοχών. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρχει παραγωγή των παρομοίων προϊόντων παντού στον κόσμο. αλλά πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Αν ένα προϊόν παράγεται απλώ μερικά χιλιόμετρα έξω από τα όρια προστασία, θα μπορούσε να βοηθήσει. Άρα δεν είναι κατά η κυρία Μακλάρκη να δούμε περαιτέρω το θέμα αλλά θεωρεί ότι μια πλήρης μελέτη αντικτύπου είναι αναγκαία πριν καταλήξουμε σε μια στρατηγική μέσο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Ο κύριος Μπίχνερ. Ως πράσινοι στηρίζουμε τη γεωγραφική ένδειξη για τα γεωργικά προϊόντα. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ελκυστική ιδέα η αρχή αυτή να επεκταθεί και σε μη γεωργικά προϊόντα για να δημιουργήσουμε για παράδειγμα σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή να διατηρήσουμε θέσει εργασία σε μια γενική περιοχή, σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά αυτό που σίγουρα δεν θέλουμε είναι το σύστημα αυτό να γίνει μια στρατηγική εμπορία των προϊόντων. Όπως έχει συμβεί με τα σήματα να κατατεθέν. Δεν θέλουμε να γίνεται κατάχρηση αυτού του συστήματος και να λέγεται για παράδειγμα ότι η μπύρα που παράγεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή τα πέτσινα σορτσάκια από το Μόναχο να μπορούν να παραχθούν πολύ μακριά από το Μόναχο. Με συγχωρείτε που αναφέρω το παράδειγμα, γιατί είναι από το Μόναχο. Όντως ισχύει όμως, ότι αυτή τη στιγμή σχεδόν κανένα πλέον βαβαρικό ε, δερμάτινο παντελονάκι δεν παράγεται στη Βαβαρία. Είμαστε διαδεθειμένοι να βοηθήσουμε ούτω ώστε να συμπεριληφθεί αυτό στι επικείμενε ανακοινώσει τη κυρία Μάλστρομ. Πρέπει να το συζητήσουμε πλήρω και θα υποβάλουμε τροπολογίε. όπου θα ορίσουμε την άποψή μα για τι αναγκαίε προποθέσει. Και θα επιμείνουμε να εκτιμήσουμε και τα μειονεκτήματα που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια νομοθετική πρόταση πριν την αποφασίσουμε. Ευχαριστώ κυρία Μπέγκη. Ευχαριστώ. Εγώ ήδη τοποθετήθηκα θετικά την τελευταία φορά που συζητήσαμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το έργο της. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο από εμπορική σκοπιά, αλλά και από τη σκοπιά της προστασίας κατά της παραποίησης. Θεωρώ και εγώ ότι μια νομοθετική δράση θα πρέπει να λυθεί σύντομα και θεωρώ άδικο να υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ της προστασίας των γεωργικών προϊόντων ε, και των ε, παραδοσιακών προϊόντων που ουσιαστικά προέρχονται από τον ίδιο οικονομικό ιστό. Αναφέρομαι, παραδείγματο χάρη, σε ορισμένε περιπτώσει όπω ε, τα μάρμαρα τη Καράρα στην Ιταλία. Δεν καταλαβαίνω γιατί και αυτό δεν θα έπρεπε να προστατευτούν με τον ίδιο τρόπο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μελέτη αντικτύπου, θα μπορούσα να συμφωνήσω. Βλέπω μικρή αναγκαιότητα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποιε θα μπορούσαν να είναι οι αντενδείξει παρά ωφέλη. Βλέπω εγώ για τους μικρούς επιχειρηματίες ε, θα θέλαμε να έχουμε ένα όσο δυνατόν πιο απλό σύστημα και όσο δυνατόν λιγότερο δαπανηρό για τις επιχειρήσεις, όμως ε, σε γενικές γραμμές υποστηρίζουμε τη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και Τζούντ. Ευχαριστώ. Συγχαίρω την Αλέσια για τη γνωμοδότηση την οποία πλήρως στηρίζω να το δω από άλλη γωνία ως Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μη γεωργικά προϊόντα όλοι θεωρούμε ότι θα ωφελούνται από προστασία γεωγραφικής ένδειξης. Και ένα το οποίο θα μπορούσα να αναφέρω είναι οι ράφτες ε, της οδού Savile Row είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, υψηλής αξίας που λειτουργούν σε παγκόσμια αγορά και συχνά αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό από ανταγωνιστές που χρησιμοποιούν ε, τον όρο Savile παρά ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη οδό. Ενδιαφέρον παράδειγμα. Γιατί στη διαβούλευση της Κομισιόν υπήρξε από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτή την περιοχή μια συμβολή όπου έλεγαν ότι οι προτάσεις για επέκταση της γεωγραφικής ένδειξης θα προστατε... προστάτευε την ε, τεχνογνωσία τους, τις δεξιότητές τους, το επίπεδο της ε, εμπειρογνωμοσύνης τους. Και τι είπαν λοιπόν στο κείμενό τους. Ε, συμμετέχοντας στη διαβούλευση για την Πράσινη Βιβλίο είπαν ότι είναι ζωτικό να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και κατάρτισής τους και να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και προστασία της αυθεντικότητας και του υψηλού επίπεδου παραγωγής. Και θεωρώ ότι όταν μια ιδέα στηρίζεται ενεργά και από τα συνδικά των εργαζόμενων και από τις επιχειρήσεις που εργάζονται, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά. Ελπίζω λοιπόν να σημειώσουμε σύντομα πρόοδο για αυτό το σημαντικό θέμα, όπως προτείνει και η συγκήτριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, παίζει ρόλο να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, λέει ο Πρόεδρος. Είμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τα συγχαρητήρια προς την εισηγήτριά μας, την Αλέσια, για τη θαυμάσια εργασία νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία, γιατί είναι ζωτική σημασία σε αυτό το θέμα, η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά προϊόντα στην εμπορική πολιτική. Το πρώτο λοιπόν είναι να αναγνωρίσουμε τη σημασία να υπάρξουν ρυθμίσεις σε ενωσιακό επίπεδο. Γιατί δεν υπάρχει ενιαία προστασία σε ενωσιακό επίπεδο. Μέλη έχουν νομοθετήματα για τα θέματα αυτά για προστασία γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί λοιπόν αυτή η κατάσταση. Βεβαίως. Από τη μία προστατεύουμε γεωργικά προϊόντα, αλλά και κάποια μη γεωργικά, όπου αναγνωρίζουμε υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος παραγωγής, ε, χειροτεχνικό σε μια συγκεκριμένη περιοχή που έχει σημαντική επίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιοχές και στην Ισπανία για παράδειγμα, σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν παρόμοια παραδείγματα, όπου ορισμένοι ζουν από ε, προϊόντα πραγματικά χειροτεχνικά, μικρομεσαίας κλίμα, ε, κλίμακας, όπου οι δεξιότητες που έχουν και προστασία που πρέπει να απολαμβάνουν είναι σημαντική και πρέπει να συνεχιστεί. Συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια ότι από εμπορικής πλευράς η προστασία των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων έχει και επιθετική και αμυντική σημασία. Είναι ουσιώδες να ληφθεί υπόψη. Η δυτή έκφραση. Και πρέπει να είναι μια δυνατότητα που θα αξιοποιήσουμε για να καταπολεμήσουμε τις απομιμήσεις και τον αθέμητο ανταγωνισμό τον οποίο υφίστανται πολλά από τα προϊόντα μας. να υπάρχει αυτή η γεωγραφική ένδειξη νομίζω ότι είναι σημαντικό για την προστασία των προϊόντων αυτών στις εμπορικές συμφωνίες που έχουμε και τις επικείμενες. Οπότε θεωρώ ότι η Κομισιόν πρέπει να υποβάλει πρόταση νομοθετική όπου αυτά τα θέματα θα λαμβάνονται πάντα υπόψη στην εμπορική μας πολιτική, στις επενδύσεις μας η προστασία αυτών των προϊόντων. Έτσι λοιπόν θα διατηρήσουμε πολλές θέσεις εργασίας και έτσι θα στηρίξουμε και τη ε, δημιουργία και νέων θέσεων εργασίας ποιότητας, σταθερές θέσεις εργασίας που θα επιτρέψουν επίσης ε, τη μείωση του πληθυσμού πολλών περιφερειών που αν δεν προστατευτούν μπορεί να καταλήξουν σε λουκέτα, μείωση ε, του πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Βαλερή Νταβινιό από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή επικρατεί τις προτάσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ιδίως ε, τη στήριξη για ένα συνεκτικό και απλό σύστημα προστασία γεωγραφικών ενδείξεων, το μη γεωργικό προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μα επιτρέψει να πετυχούμε αντίστοιχα επίπεδα προστασία μη γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων, αλλά και σε πολυμερέ επίπεδο. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμα αποφασίσει να δώσει συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία, όμως Κατά τη λήψη απόφαση ε, για το πώ θα κινηθούμε περαιτέρω σε αυτό το φάκελο, θα λάβουμε υπόψη ω Κομισιόν τι προτάσει τη ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να αποφύγουμε περιττή γραφειοκρατία, μείωση των ε, προτύπων ασφαλείας που ήδη υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη και μετά τις, ε, τη θετική ανταπόκριση της Επιτροπής Γεωργικών Υποθέσεων και τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών και τη ΝΕΟΚΕ, η πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου θα βοηθήσει να θα συγκαθορίσει μάλλον τη συνέχεια που θα δοθεί στο έργο μας. Ευχαριστώ. Η Αλέσια. Ευχαριστώ. Εγώ άκουσα τα διάφορα σχόλια και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η απάντηση σε ορισμένε από τι ανησυχίε που προέκυψαν ε, από τι παρεμβάσει των συναδέλφων είναι εξή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτή η πρωτοβουλία, η γνωμοδότηση που παρουσιάζουμε για την πρωτοβουλία αυτή, έχει ω θεμελιώδε πυλώνε κάποια από τα θέματα αξιακά που προέκυψαν ε, στις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων. Και κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν για να βρούμε και τους πρακτικούς τρόπους και τα πρακτικά μέσα μέσω των οποίων θα έχουμε στην δυνατόν πιο αποτελεσματική γνωμοδότηση. Μία τέτοια πρωτοβουλία χρησιμεύει για να προστατεύσει, να ενισχύσει και να αξιοποιήσει όλη την πολιτιστική και οικονομική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμεύει για να ενισχύσει την ικανότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεών μας. Ε, έτσι λοιπόν ε, θα έχουμε και προσθέτει αξία, οικονομικά ωφέλη και όλα αυτά θα αξιοποιήσουν την κληρονομιά ε, των γνώσεων, των εμπειριών, των αρμοδιοτήτων και ε, κάποιες ε, ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος μέσω του οποίου εμείς μπορούμε να αποφύγουμε να τοποθετηθούμε είτε να τοποθετηθούμε με τρόπο μη στρεβλωτικό σε σχέση με τον τελικό μας στόχο. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε κατά νου τις αξίες αυτές και αν κατορθώσουμε με την έκθεση αυτή να εντοπίσουμε όλες τις δυνατότητες που ενέχονται στις σχέσεις με τις ε, τρύπες, τρίτες χώρες, τότε δεν θα πρέπει να ανησυχούμε. Και εγώ νομίζω ότι η φιλοδοξία μας θα πρέπει να είναι η εξή να ζητήσουμε να υπάρχει ως δυνατόν πιο συνεκτική ρύθμιση και να μην υπάρχουν επικαλύψεις με τα εφιστάμενα. Γιατί εγώ νομίζω ότι δεν θα προσφέρουμε καλή υπηρεσία και δεν θα εξυπηρετήσουμε τους στόχους που έχουμε διαφορετικά το αντίθετο μάλιστα θα έχουμε επιβάρυνση της νομοθεσίας, κάτι που δεν είναι στις προθέσεις μας. Ε, ακριβώς, να το προσέξουμε αυτό. Προθεσμία για τροπολογίες 11 Μαΐου, 5 ώρα το απόγευμα. Και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε την έκθεση τον Ιούνιο. Οπότε λύγει το δημόσιο τμήμα της ε, συνεδρίασής μας και σε δύο λεπτά θα έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών.